Κυρίες και κύριοι, είναι απαραίτητο νομίζω να ξεκινήσουμε. Δεν μπορούμε εμείς που ερχόμαστε στην ώρα μας να ε, φέρουμε και την ευθύνη για όσους έχουν καθυστερήσει και να υφιστάμε αυτές τις συνέπειες. Yeah, Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir setzen unsere Sitzung fort. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίαση αγαπητοί συνάδελφοι με το σημείο 23 της ημερήσιας διαταξής. Μετά το μαραθώνιο των ψηφοφοριών πάλι θα συζητήσουμε τώρα θέματα ουσίας. Έχουμε ε, σημαντικές προσωπικότητες εδώ προσκεκλημένες που θα μας δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και ελπίζουμε να έρθουν και αρκετοί συνάδελφοι. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση της τελικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ασφάλειας της Έρευνας και της Καινοτομίας. Καλωσορίζω εδώ τον κύριο Μάτε, Δράγμουτιν Μάτε, πρόεδρο του κέντρου, του ΕΣΤΡΙΦ. Καλωσορίζω και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να μπορούμε και από τις δύο πλευρές να ρίξουμε φως στην υπόθεση αυτή. Παρακαλώ, κύριε Μάτεν. Ας μην καθυστερήσουμε πρώτα. Mogoče najprej dve, tri besede v mojem jeziku. Eh, lepo pozdravljeni, eh, gospod predsednik. Ε, να πω λίγα πράγματα στα σλοβενικά για να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, παρουσίαση. Αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής Ήτρε, χαίρομαι που μπορώ να βρίσκομαι εδώ και να σας απευθύνω το λόγο εξ ονόματος της ΕΣΡΙΦ, να σας παρουσιάσω και τι έχουμε κάνει μέχρι τούδε. Έχουμε προσκομίσει και υλικό το οποίο μπορείτε να διαβάσετε αργότερα και τώρα θα συνεχίσω στην αγγλική, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολα για όλους. Η ΕΣΡΙΦ ε, περιλαμβάνει περίπου 46 μέλη της Ολομέλειας από 31 ε, χώρες ε, και έχουμε εκπροσώπους της βιομηχανίας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά Ινστιτούτα, πανεπιστήμια, καθώς επίσης και μη κυβερνητικού οργανισμούς και οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πάνω από 600 εμπειρογνώμονε, οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο της ΕΣΡΙΦ μέσω 11 ομάδων εργασία. Αυτό είναι μία μοναδική διαδικασία μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργαζόμαστε εδώ και δύο χρόνια. Και τι έχουμε κάνει σε αυτά τα δύο χρόνια. Ασχολούμαστε με θέματα ασφαλείας και θέλουμε να συνεισφέρουμε σε μία πιο ασφαλή Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη να βρούμε ε, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποδοτικά όλες μας τις πηγές, ε, τι, έχουμε, τι στοιχεία έχουμε από την καινοτομία και την έρευνα και να συμπεριλαμβάνουμε και αυτά τα αποτελέσματα στην ε, πολιτική βιομηχανίας. Και έτσι θα μπορέσουμε να κλείσουμε και ένα κύκλο με τους τελικούς χρήστες. Η βιομηχανία θα πρέπει να μας παρέχει τον καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια. Σε αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε μέσω της δουλειά μα να βρούμε τις απαντήσεις στον τομέα της καινοτομία, της έρευνα και της βιομηχανία. και να φροντίσουμε ώστε να μην ε, προσβάλλονται οι αξίε μα με κανένα τρόπο. Η κοινωνία μα εξαρτάται από την τεχνολογία και τι υποδομέ, όπω για παράδειγμα τα δίκτυα ηλεκτροδότηση, το διαδίκτυο, τι δημόσιε μεταφορέ, την αεροπλοεία, τι τηλεπικοινωνίε κ.ο.κ με μικρή προσπάθεια είναι σε γενικές γραμμές εύκολο να διαταραχθούν όλες αυτές οι υποδομές από τις οποίες εξαρτώμεθα στην καθημερινή μας ζωή. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ταυτόχρονα και τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν και την ασφάλειά μας ε, έξωθεν. Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις και πολλές περισσότερες. Οι απαντήσεις μας είναι οι εξής. Θα πρέπει να έχουμε βασικά μηνύματα, συστάσεις και ε, μία ατζέντα ευρωπαϊκής ε, έρευνας και καινοτομίας για την ασφάλεια. Ε, η ΕΣΡΙΒ εντόπισε αρκετούς τομείς στους οποίους πρέπει να έχουμε βασικές δυνατότητες και δυνατότητα έρευνας και τα διαχωρίζουμε αυτά σε πέντε κλάδους. Έχουμε ένας κύκλος ασφάλειας για την πρόληψη, την προστασία, την προετοιμασία, την, ε, την ανταπόκριση και την ανάκτηση. Εστιάζουμε κυρίως στην ασφάλεια των ανθρώπων. Ο δεύτερος ε, πυλώνας ε, ασχολείται με τα διάφορα μέσα επίθεσης που μπορεί να έχουμε, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένους και προβαλόμενους μελλοντικού κινδύνους και εξετάζουμε τρόπους για να ανεχνεύσουμε ε, συμβατικές και μη συμβατικές επιθέσεις. Ο τρίτος πυλώνας ασχολείται με τα κρίσιμα σημεία ασφάλειας, όπως για παράδειγμα η ενέργεια, οι μεταφορές και άλλες κρίσιμες υποδομές, όπως για παράδειγμα η διασφάλιση της ύπαρξης βασικών δυνανοτήτων ε, κατασκευή στην Ευρώπη. Ο τέταρτος πυλώνας θέλει να διασφαλίσει την ταυτότητα, την πρόσβαση και την μετακίνηση των ανθρώπων και αγαθών. Κυρίως εστιάζει στην ασφάλεια των συνόρων και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έχουμε ε, ασφαλή διαχείριση ταυτότητας. Ο τελευταίος πυλώνας ασχολείται με εγκάρσιας δυνατότητες Και η ασφάλεια αφορά και το ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα διαστήματος. Η ατζέντα αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί με κάποιες βασικές αρχές. Οι βασικές αρχές αυτές ε, παρουσιάζονται στα βασικά μας μηνύματα και μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες της κοινωνίας και τις ατομικές μας ελευθερίες. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε απολύτως τον κάθε ε, υπαρκτό και άγνωστο κίνδυνο που έχουμε για το μέλλον, αλλά πρέπει να έχουμε στεναρή προστασία από τους σαφείς και παρόντες κινδύνους. Επίσης πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία μας για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των γνωστών κινδύνων και το κοινό κατανοεί ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Αλλά θα ήταν απαράδεκτο να μην είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε γρήγορα και αποτελεσματικά ε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ο στόχος λοιπόν είναι να έχουμε κοινοτική ανοχή. Ε, τα βασικά στοιχεία είναι να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ κοινού και των ε, ε, αρχών διακυβέρνησης και αυτό το επιτεχάνουμε μέσω διαλειτουργικότητα σε όλες τις πτυχέ. Τα ωφέλη της νέας τεχνολογίας, τα οποία αναπτύχονται σε μια συστημική προσέγγιση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μα σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι οργανώσεις που ασχολούνται με τα καταπήγοντα θέματα ε, θα έχουν τη δυνατότητα να ε, είναι διαλειτουργικές, να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση και επίσης οι πολίτες θα πρέπει να ε, εξοικειώνονται ακόμα περισσότερο και να γνωρίζουν τα επίπεδα διαφάνειας ε, της επικοινωνίας και του σχεδιασμού που σχετίζονται με την ασφάλεια. Και εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικές βιομηχανικές δυνατότητες και μία βάση γνώσεων, αλλά είναι μία κατακαιρματισμένη αγορά ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνουν κοινέ προσπάθειες για να έχουμε περισσότερη ευρωπαϊκή ασφάλεια η οποία θα ε, υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή πολιτική Αυτή η πολιτική βιομηχανία θα πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία και ταυτόχρονα η ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθεί ε, στα ε, προκαταρκτικά στάδια προγραμματισμού. Στην έκθεσή μας κάνουμε και κάποιες συστάσεις για να έχουμε υψηλότερες ε, έρευνες και αποτελέσματα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας για την ασφάλεια. Οι συστάσεις συμπεριλαμβάνουν κοινέ ευρωπαϊκές δυνατότητες, νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, καθώς επίσης και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια, την παγκόσμια διάσταση και το μέλλον της ε, έρευνας για την ασφάλεια. Να σταθώ σε μία από τις πολλές μας συστάσεις. Η ΕΣΡΙΑ προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει το παρόν καθεστώς ε, ανάπτυξης ε, για τα ερευνητικά προγράμματα ασφάλειας με στόχο να έχουμε ένα ετήσιο προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τα εθνικά προγράμματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και αυτό το βαθμό φιλοδοξίας. Να σας δώσω μια πολύ σύντομη εικόνα των κυρίων συμπερασμάτων που έχει εξαγάγει η ΕΣΡΙΒ. Για Σας έχει δοθεί μία σύντομη ε, σύνοψη. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει περίπου 40 σελίδες και αναφέρει διεξοδικά τα στοιχεία τα οποία σας παρουσίασα και υπάρχει και μία σύντομη σύνοψη της δουλειάς μας και στο δεύτερο μέρος έχουμε πάνω από 250 σελίδες ε, κειμένου από κάθε ομάδα εργασίας από τις 11 που έχουμε. Η κάθε ομάδα εργασίας έχει ένα δικό της ε, τμήμα αφιερωμένο ε, σε αυτήν ειδικά στην έκθεση και εκεί θα βρείτε τα στοιχεία για την έρευνα καθώς επίσης και πολύ ενδελεχή προγράμματα για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης για το μέλλον και ένας πίνακας για την έρευνα και τις προτεραιότητες που θέλουμε να έχουμε στην έρευνα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας την παρουσίασή μου, να πω ότι η Έσριφ προσπάθησε να βρει πολύπλοκες απαντήσεις, διότι έχουμε πολύ πολύπλοκα ερωτήματα. Θεωρούμε ότι με αυτή την έκθεση δίνουμε κάποιες απαντήσεις για όσους λαμβάνουν αποφάσεις, για τους πολιτικούς σε όλα τα επίπεδα, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το Συμβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και για, τον, ε, για τη βιομηχανία στην Ευρώπη και για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Ελπίζω να διαβάσετε την έκθεση και να βρείτε και την πλειονότητα των απαντήσεων σε αυτά που αναζητάτε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Äh, Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και αν συμφωνείτε Καταρχήν θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση και ο κύριος Βάιζενμπέργκερ αντιλαμβάνουμε δεν είναι εδώ αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριος Μαλανκάρνε ελπίζω ότι δεν ε, έχω προφέρει λάθος, το όνομά του. Θα ήθελα πάντως να του δώσω το λόγο για να μπορέσει να μας παρουσιάσει ε, τα σχόλιά του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται στις υπηρεσίες και στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ε, καταρτίστηκε από διάφορες υπηρεσίες. Δεν θα αναφερθώ λοιπόν σε όλα τα θέματα τα οποία έφυξε η έκθεση, ε, απλώς θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Καταρχήν θα ήθελα να επενέσω την πολύ σημαντική εργασία η οποία έγινε ε, γιατί όλα τα κράτη-μέλη έχουν νέους τομείς έρευνας και έτσι τώρα είμαστε στο τρίτο έτος της εφαρμογής του προγράμματος ερεύνης και ε, παρόλο που έχουμε ένα ποσοστό επιτυχίας 1 ε, ε, στα 5, νομίζω ότι προχωρούμε καλά και υπάρχει και το θέμα της έρευνας. Διαπιστώνουμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε την τεχνολογία με τις ανάγκες της κοινωνίας διότι αυτό είναι κάτι που παρουσιάζεται όλο και πιο έντονα αν δούμε το παράδειγμα των τεχνολογιών που αναφύνονται στους αρωτές σώματος ή σε ε, άλλες ε, τεχνολογίες για ε, λύσεις ασφαλείας που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Δεύτερον, θα θέλαμε να υποφεληθούμε της πολύ χρήσιμης ε, ε, συμβουλής ε, όσον αφορά την εσωτερική πολιτική διότι η βιομηχανία δεν έχει, δεν έχει διευκρινιστεί δηλαδή ποιοι είναι οι διάφοροι τομείς έχουμε κάνει μια πρώτη χαρτογράφηση αλλά όλα αυτά πρέπει να συνεχιστούν και θα χρειαστεί να βρούμε μέτρα για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Πέραν αυτών των δύο διαστάσεων θα ήθελα να αναφέρω ότι κάτι το οποίο ίσως είναι αντιφατικό. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ε, οι ηθικές προδιαγραφές ε, πέραν των τεχνικών προδιαγραφών και θα έπρεπε να τις συνδυάσουμε. Ε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την σήμανση και τότε ίσως η βιομηχανία θα μπορούσε να είναι πολύ ανταγωνιστική αλλά είναι μια πρώτη παρατήρηση και θα περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας για να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ θερμά και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που το επιθυμούν, καταρχήν στον Κριστιαν Έλερ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους διότι είχα παρακολουθήσει κοινοβουλευτικά και συνοδεύσει την διαδικασία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ΕΣΡΙΦ προσπάθησα δηλαδή του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ασφαλείας ακόμη και αν ήμουνα στο Στρασβούργο ο Μάρτιν προσπάθησε όντως να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και όταν πια το θέμα λειτουργούσε και υπήρχαν 600 ερευνητές και αστυνόμοι, εκπρόσωποι των πνευματικών επιστημών όταν δηλαδή υπήρχε μία πολύ εκτενής προσπάθεια και την οποία έπρεπε να ολοκληρώσουμε ε, νομίζω ότι μπορέσαμε να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά ε, και ότι ανταποκριθήκαμε στις προσμονές. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή που υπήρξε θαραλέα. Η Επιτροπή δεν είναι συνήθως τόσο ειλικρινή σε μια τέτοια συζήτηση, διότι όταν έχουμε 600 προσωπικότητες που ερωτούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη επί δύο χρόνια, ε, έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις. Ε, ε, και ξεχνάμε ποιους έχουμε ερωτήσει και ποιους όχι. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή έκανε εξαιρετική δουλειά διότι η έκθεση αυτή μας δίνει μία προοπτική η οποία αναφέρεται στην ευρωπαϊκή διάρθρωση ασφαλείας και είναι άλλωστε μία προοπτική για μία εικοσαετία. Ε, το τρίτο θέμα είναι το κατά πόσον το θέμα είναι επίκαιρο διότι ξέρω ότι το θέμα είναι περίπλοκο αλλά θα ήθελα να αναφέρω μερικούς αριθμούς για να δείξω πόσο σημαντική είναι, αυτή, ε, είναι αυτό το θέμα. Σημαντική δεν είναι μόνο η έρευνα, αυτό που είναι σημαντικό είναι οι ε, δύο, οι δύο ε, διακοπές ηλεκτρικής παροχής που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη όπου ε, δεν υπήρξε πλέον παροχή ρεύματος στη μισή Ευρώπη μας απέδειξε ότι μπορεί να έχουμε μια εσωτερική αγορά μπορεί να έχουμε αγωγημότητα αλλά πέραν αυτών πρέπει να προχωρήσουμε πάμε πέραν των βάσεων της κοινωνίας της Ευρώπης διότι δεν προσπαθούμε να εξετάσουμε ένα εξατικό, εξωτικό ερευνητικό θέμα και εδώ δεν μιλώ πλέον για τρομοκρατία αναφέρομαι σε ε, δύο πολύ απλά παραδείγματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που οδήγησαν σε τεράστια προβλήματα. Μετά, η κοινή αγορά. Ε, το θέμα της ε, ερεύνης δεν τίθεται απλά. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε με την ε, πολιτική ε, βιομηχανικής πολιτικής διότι η αγορά αυξάνεται ε, κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι από εκεί που είχαμε μία αγορά 2 δισεκατομμυρίων ευρώ τώρα έχουμε μία αγορά των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναπτύσσεται και να αναπτύσσεται διεθνώς. Δηλαδή το θέμα της ασφαλείας και η έρευνα στον τομέα της ασφαλείας δεν είναι μόνο θέμα ερευνητικό αλλά είναι και θέμα επιβιώσεως της βιομηχανίας της Ευρώπης και ε, επίσης το θέμα της ε, έρευνας ε, στην Ευρώπη είναι μια ανομαλία διότι πλέον ε, δεν μιλάμε μόνο για μια αρχιτεκτονική ασφαλείας ε, διότι δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε πολιτικά. Είχαμε λοιπόν συμφωνήσει να γίνει ένα τεράστιο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο τότε κάλυπτε από 230 εκατομμύρια στο, και αυξήθηκε στο ποσό του 1,4 δισεκατομμύρια και αυτό μέσω της παρεμβολής του Κοινοβουλίου το οποίο επέμεινε ότι χρειαζόμαστε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τότε λοιπόν ανακοίνωσε για πρώτη φορά το Συμβούλιο μία ε, μελέτη για μια ευρωπαϊκή διάρθρωση ασφαλείας. Έχουμε εδώ πάρα πολλά εργαλεία, πάρα πολλές δηλώσεις για μελλοντικά σενάρια και ε, θα έπρεπε να δούμε αν μπορούμε πλέον να συζητάμε για μια αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη και αν η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφωνούν σχετικά με αυτό το θέμα ή όχι, διότι είναι προφανές ότι θέλουμε να υπάρχει έρευνα στο μέλλον, αλλά καταρχήν στην έκθεση που καταρτίστηκε θα έπρεπε να καθορίσουμε ποια είναι τα κεντρικά θέματα που έπρεπε να απασχολήσουν την έρευνα στην Ευρώπη. Και υπήρξε ένας κατάλογος Μοναδικό μοναδικός 600 ε, ε, οργάνων από όλες τις χώρες ένα πολύ περίπλοκο θέμα το οποίο προφανώς ε, έχει και ορισμένες ελλείψεις αλλά μας έδωσε μία πρώτη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα πολιτικά δεδομένα βάσει αξιοπίστων επιστημονικών σεναρίων. Δηλαδή ε, ξεπεράσαμε την ε, πολιτική της έρευνας και συγχρόνως ε, ξεκινούμε να συζητάμε τις ευρωπαϊκές δομές ασφαλείας και ε, υπήρξαν και επιστημονικές επιπτώσεις και πέραν αυτού το ερώτημα του πόσο ασφαλής είναι η δομή της κοινωνίας της Ευρώπης η οποία ε, πρώτη φορά παρουσίασε τέτοια θεματολογία. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να διαβάσουμε την εκτελεστική έκθεση σαν Γερμανός θεωρώ πάντοτε ότι ε, έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της κοινότητας και πολύ λυπούμε ότι υπάρχει μόνο αγγλικά και γαλλικά και ήθελα να το δω και γερμανικά και υποθέτω και ιταλικά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει γιατί δεν πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό απλώς σαν ερευνητικό αλλά σαν ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ και στο μέλλον. Και μία τελευταία φράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι οι νέες συμφωνίες ζητούν να υπάρξουν και νέα ε, καθήκοντα, ε, ποιες είναι οι σχέσεις με την άμυνα, ε, τι γίνεται με τις εξωτερικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι συμβαίνει με την αντιμετώπιση των καταστροφών, των φυσικών καταστροφών. Στο παρελθόν ήμασταν πάρα πολύ ευέλικτοι στα θέματα αυτά. Αλλά η δήλωση ε, την οποία ακούω αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ε, μία preparatory action, δηλαδή ε, μία προκαταρκτική δράση για να ερευνήσει τα αμυντικά θέματα επί των οποίων μέχρι στιγμής δεν υπήρχε συμφωνία. Οπότε πρέπει να δούμε αν έχουν διαφανεί κάποιες λύσεις ή αν πρόκειται πρόκειται ε, να προχωρήσουμε στα θέματα της αμυντικής έρευνας, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαντουρέλα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πολύ σύντομα θα ήθελα να πω στον κύριο Μπότ Μάτε εξ ονόματο τη ομάδα μα την ικανοποίησή μα για την παρουσίασή του εδώ και να τον ευχαριστήσω για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μα έκανε για το έργο του οργανισμού που εκπροσωπεί. Ο τομέας της ασφάλειας είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός, τομέας προτεραιότητας στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και νομίζω ότι είναι ένας από τους εννέα τομείς που επιλέχθηκαν τελικώς για το 7ο πρόγραμμα ε, πλαίσιο σε θέματα συνεργασίας και όπως είπατε πολύ σωστά και εσάς και εσείς ο τομέας της ασφάλειας επιδρά πολύ σημαντικά στους πολίτες, διότι όλοι θέλουμε μια πιο ασφαλή Ευρώπη και είναι και ένας από τους πιο άγνωστους ε, τομείς, αυτούς που δεν γνωρίζουμε και τόσο καλά και έχουμε συζητήσει λιγότερο εδώ στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό ακριβώς σας ευχαριστώ διπλά για την παρουσία σας εδώ γιατί αποτελέσατε και το έναυσμα για πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από τους συναδέλφους. Από τα όσα μας είπατε για την ΕΣΡΙΦ θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πράγματα και να σας ρωτήσω ε, ως χρήστη του 7ου προγράμματος πλαίσιο θα ήθελα να ξέρω πώς λειτουργεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στο δικό σας τον τομέα διότι όπως πολύ σωστά είπε και ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρισκόμαστε πλέον ε, στα μισά του δρόμου και θα πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση οι προτάσεις σας θα μπορούσαν να είναι πολύ ενδιαφέρουσες ε, διότι θέλουμε να προετοιμάσουμε και το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι τα πράγματα τα οποία θα αλλάζατε εσείς, ποια είναι πράγματα θα θεωρείτε ότι χρήζουν βελτίωση στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία ε, να μιλήσετε και σλοβενικά. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου πρόταση και εμένα, λέει η κυρία Ζόρνταν Σίζελ. Και το εννοώ. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τους δύο προσκεκλημένου για τις παρουσιάσεις τους, ιδιαίτερα τον κύριο Μάτε, διότι με μεγάλη χαρά ακούω να μιλάει κανεί στην Επιτροπή μας σλοβενικά Και ειδικά όταν ε, πρόκειται για μια προσωπικότητα τόσο διακεκριμένη, τον κύριο Μάτε, πρώην Υπουργό Αμήνης. Μεγάλη λοιπόν ε, η σημασία της παρουσίας σας. Πρέπει να πω ότι εγώ μόνο τη συνοπτική έκδοση είδα, στις τέσσερις σελίδες, έτσι έχω μόνο πολύ γενικές ερωτήσεις, δύο τον αριθμό. Είχαμε κάποια προγράμματα μέχρι τώρα, προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν από την προηγούμενη εντολή και προσπαθούμε τώρα να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν σε διάφορα επίπεδα τα προγράμματα αυτά. Πιστεύω δε ότι υπάρχει διαφορά ως προς την υλοποίηση των προγραμμάτων ανάλογα με τον αριθμό των μελών των ομάδων που θα συμμετάσχουν τη κάθε ομάδα που συμμετάσχει στα προγράμματα αυτά. Αυτό εδώ ακριβώ εντοπίζω το εγώ το πρόβλημα, γιατί πρέπει να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να αναπτύσσεται ομοιογενώ, όχι με διαφορετικέ ταχύτητε. Πρέπει όλοι οι πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ισότιμη πρόσβαση. Και γι' αυτό από εσά θα ήθελα να ακούσω τι είδου συστάσει έχετε να προτείνετε, έτσι ώστε η ασφάλεια, η έρευνα για την ασφάλεια, να είναι κατά ισότιμο τρόπο ε, ανοιχτή σε όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες στα προγράμματα αυτά. Μια άλλη ερώτηση. Προδιαγραφές ειδικέ, προδιαγραφές δηλαδή όπως αυτή τη προστασία προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει ασφαλώς να λαμβάνονται υπόψη στην ε, έρευνα για την ασφάλεια, η οποία γνωρίζουμε ότι αποτελεί και μια καλή βάση για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ε, βιομηχανίας μας. Ως εκ του λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε τι ε, θα βλέπατε ως βέλτιστη λύση ε, για να εκφραστούν όλα αυτά σε, μια πρακτική, σε ένα πρακτικό σύστημα. Ευχαριστώ. Κύριος Κοραρδεκάμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάτε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεσή του και θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης και για τη συνοπτική ε, μορφή του βιβλίου που εκφράζει και τις βασικές γραμμές της φιλοσοφίας του, της φιλοσοφίας ως προς την ασφάλεια. Ερωτήσεις λοιπόν, πρώτη. Ποιος ορίζει τους βασικούς άξονες τις ε, βασικές δηλαδή απειλές. Ποιος τους ορίζει, ποιος τις ορίζει. Κάποιος από την Επιτροπή, κάποιος υπεύθυνος του τέταρτου λεγόμενου πυλώνα, το φόρουμ το ίδιο. Θα είναι εκείνο το οποίο θα προσδιορίσει, το έστριφλε το ίδιο, θα προσδιορίσει ποια είναι αυτή η νέα απειλή. Και άλλη μία απλή και πρακτική ερώτηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με το κινητό τηλέφωνο ε, είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους ασφαλείας, υποκλοπές κτλ. Οι αρχές λοιπόν, οι θεσμικές αρχές των κρατών ενδέχεται και να εξασφαλίσουν την άδεια για παρακολούθηση των συνδιαλέξεών μας. Ναι. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες θα επέτρεπαν στον καθένα να υποκλέψει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις χωρίς την παραμικρή άδεια του συνδιαλεγωμένου. Ξέρω ότι υπάρχουν και πλέον ε, στην αγορά μικρόφωνα ε, τα οποία από απόσταση μπορούν να πιάσουν τους ήχους μιας Έρα το λοιπόν. Εάν το ΕΣΡΙΦ θεωρεί ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο ασφάλεια, δηλαδή η πιθανή προσβολή των ανθρωπινών δικαιωμάτων, των ατομικών δικαιωμάτων αποτελεί κίνδυνο ασφάλεια. Γιατί το πρόβλημα εδώ δεν είναι η τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει αυτή την παραβίαση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και η τεχνολογία η οποία επιτρέπει να αντιμετωπιστεί η παραβίαση, να αποτραπεί δηλαδή. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ καταρχά συγγνώμη που έφτασα με καθυστέρηση. Κύριε Μάτε και κύριε εκπρόσωπε τη Επιτροπή, με συγχωρείτε. Έχω μια απλή και πρακτική ερώτηση Ξέρετε ότι είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες την ψηφοφορία για τη συμφωνία SWIFT με τις ΗΠΑ, τη συστήσαμε διεξοδικά και εν τέλει την απορρίψαμε. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσει σε νέα διαπραγμάτευση. Μέσα στη συζήτηση λοιπόν εκείνη, το διαρκώ το ζήτημα το κατά πόσον η Ευρώπη είναι σε θέση να ε, εξασφαλίσει αυτό το οποίο μπορούν να έχουν οι Αμερικανοί τώρα ήδη με την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του SWIFT μέσω ενός βελγικού σερβερ, εξυπηρετητή. Ε, ερωτώ λοιπόν εάν η Ευρώπη, όχι τώρα φυσικά, αλλά γενικά ε, σαν ε, θεωρία μπορεί, με ποιου όρου, με ποιο κόστος, με ποιο σύστημα να αναπτύξει δυνατότητε πρόσβασης αντίστοιχε με αυτέ που έχουν οι Αμερικανοί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σένσου παρακαλώ, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, ομιλίες σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δραστηριότητα του Έστριφ που μας ε, παρουσιάσατε. Βλέπω ότι είναι η πρώτη φορά που ενημερώνομαι τόσο διεξοδικά για τις δραστηριότητες του φόρουμ σας και θα ήθελα αφενός με να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου και να κάνω ένα σύντομο σχόλιο μας με μια ερώτηση. Πώς ενημερώνετε τους θεσμούς, τις αρχές στα κράτη-μέλη για τα πορίσματα των δραστηριοτήτων των σας. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε για να παρακολουθήσετε εάν όντως τηρούνται ή σε ποιο βαθμό τηρούνται οι συστάσεις σας από την Ένωση και τα κράτη-μέλη για τα ζητήματα της ασφάλειας. Και επίσης έχω άλλη μια ερώτηση. Συναφεί και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πατρίδας μου, της Ρουμανίας. Ξέρω ότι έχετε αναλάβει στην τελευταία περίοδο κάποιες μελέτες ε, και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε εκπονήσει μελέτη σχετική με την δυνατότητα πρόβλεψης σεισμού Ξέρετε ότι η Ρουμανία τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί επανειλημμένως από σεισμικές διονύσεις. Βρισκόμαστε σε μια ε, περιοχή ιδιαίτερα σεισμογενή και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω αν έχετε κάποια στοιχεία. Και εν τέλει, την πλήρη έκδοση της έκθεσής σας, πού μπορούμε να τη βρούμε. Είπα, έχετε κάποια ιστοσελίδα στην οποία μπορούμε να τη διαβάσουμε, μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάνη Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις πληροφορίες, για την ενημέρωση που μας δεθέσατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις λοιπόν. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και πού εντοπίζετε τα νευραλγικά σημεία του ε, έργου σας. Ασφαλώς ε, θα υπάρχουν κάποιες περιφέρειες ή κάποιοι θεσμοί, κάποιες αρχές που θεωρείται πιο κεντρικής σημασίας. Ε, ίσως υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία εντοπίζετε τους εγκεφάλους εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν ε, τα επόμενα 20 χρόνια Φερπίν να μας ε, προσφέρουν αποτελέσματα συγκεκριμένα από τη δουλειά τους. Και βεβαίω έχουμε και το ίντερνετ, έχουμε την ψηφιακή ατζέντα, ψηφιακό πρόγραμμα, το οποίο έχει αναχθεί πλέον ε, σε μεγάλη σημασία θέμα και έχει αποτελέσει ειδικό χαρτοκυφυλάκιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ με στην έκθεση δεν βλέπω γιατί πράγμα ακριβώς γίνεται λόγος στις απειλές που καταγράφονται ως προς το ίντερνετ, παραδείγματι. Είχαμε μια επίθεση μέσω του ίντερνετ τα τελευταία χρόνια. Τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα, μπορείτε να δώσετε κάποιες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο κύριος Μέσαρος. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Μάτε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Οι στόχοι και τα οράματα τα οποία μας περιγράψατε είναι ύψης της σημασίας και εγώ προσωπικώς έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια είναι τα μέσα, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία αξιοποιείτε στην έρευνά σας. Γιατί είναι μια ιδιάουσας μορφής έρευνα, μια ξεχωριστή έρευνα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε εδώ κάποια πρότυπα ή προσωμιώσεις, ενδεχομένως μέσω του ίντερνετ. Έχετε στηριχθεί για την έρευνά σας σε επιστημονικές υποθέσεις και πιθανές ε, ε λύσεις. Ευχαριστώ και σύντομα ο κύριος Έλλερς. παρακαλώ για να κλείσουμε. Κρίστιαν, ήθελες κάτι ακόμα να πεις έτσι, δεν Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση ακόμη διότι ε, ακούσαμε πολλές ε, προτάσεις, συστάσεις αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σκέφτεται ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή θα υπάρξει κάποια ε, δομή, υπάρχουν ε, προκαταρκτικές συζητήσεις για ένα πρόγραμμα πλαίσιο 8, ε, υπάρχουν συμπεράσματα τα οποία θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποιο σημείο βρίσκονται όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και μετά ε, με το θέμα που ανέφερε ο συναδερφός διότι το Κοινοβούλιο ε, έχει πάρα πολλές ερωτήσεις. Μιλάμε όλοι για ε, δοκιμασίες ασφαλείας, για το κυβερνο, ε, το έγκλημα στο διάστημα. Υπάρχουν διάφορα θέματα και ε, το υπεύθυνο γραφείο η Ενίσα βρίσκεται στο Ηράκλειο στην Κρήτη και ε, έχει ε, ένα προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων για να πληρώνει το προσωπικό και ε, να μπορεί να καταρτίζει ένα-δύο προγράμματα το χρόνο. Το ερώτημα είναι εάν μπορούν τα προγράμματα αυτά να εφαρμοστούν ή αν όλη αυτή η αν όλοι είναι χωρίς αποτέλεσμα. Ε, δεν έχει να κάνει κάτι με το κράτος μέλος αυτό, αλλά η ενίσα αυτή τη στιγμή ε, έχει ε, μία σύνδεση με την οποία μπορεί να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία μόνο διότι δεν υπάρχει καλή ε, σύνδεση στο διαδίκτυο, ε, παροχή ίντερνετ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για πάρα πολλά προβλήματα που μας απασχολούν ε, και υπάρχει ένα ευρωπαϊκό γραφείο το οποίο βάλαμε σε ένα ελληνικό νησί που δεν έχει σύνδεση με το ίντερνετ και χρειάζεται 8 ώρες για να έρθει κάποιος αεροπορικός από εκεί έως τις Βρυξέλλες και για λόγους κόστους ο, εκπρόσωπος μπορεί μόνο να ταξιδέψει με ορισμένες συνδέσεις. Αυτή είναι ασφάλεια για τα εγκλήματα στο κυβερνοχώρο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν υπάρχει κανένα νόημα να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε αυτή την εταιρεία. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ξέρω εάν μπορείτε τώρα να προσπαθήσετε να απαντήσετε. ο συνάδελφος ο κύριος Τσίζελ μου θύμισε ότι έρχομαι από ένα μικρό κράτος οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω στη γλώσσα μου. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι η έκθεσή μου δεν περιείχε περισσότερες λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να απαντήσω σε ερωτήματα που είχατε θέσει αλλά πρέπει να σας πω ότι ο χρόνος που είχα για να ετοιμάσω αυτή την πρώτη παρουσίαση ήταν πολύ περιορισμένος. Η ΕΣΡΙΦ ε, ουσιαστικά δεν προβαίνει σε έρευνα αυτή καθεαυτή. Απλώς συγκεντρώνει όλα τα κράτη-μέλη, όλα τα ευρωπαϊκά γραφεία στον τομέα της ασφαλείας και ο κύριος Σέλερ όπως είπε ήταν μέλος της ΕΣΡΙΦ και συγχρόνως εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαφόρων εταιριών, οργάνων ε, έρευνας, οργανισμών έρευνας, δηλαδή είχαμε 64 μέλη ε, εις ε, το Ευρωπαϊκό αυτό φόρουμ για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ασφάλειας, τα οποία είχαν επιλεγεί δια και αποφάσιζαν δια Και η τελική έκθεση είναι το αποτέλεσμα συνενέσεως ε, μεταξύ των ε, διαφόρων εμπλεκομένων. Είχαμε 11 ομάδες εργασίες οι οποίες ασχολούνται με διάφορα θέματα και νομίζω ότι η μεγαλύτερη προτιθέμενη αξία για τις έρευνες που κάνει το φόρουμ αυτό είναι ότι δεν επικεντρωθήκαμε μόνο στις τεχνικές λύσεις σχετικά με την ασφάλεια των αεροδρομίων, την ασφάλεια των συνόρων, ε, ε, αλλά για πρώτη φορά ε, συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να εμπλακεί στην έρευνά μας και ένα στοιχείο κοινωνιολογίας, δηλαδή ότι χρειαζόμασταν κοινωνική ανοχή αντοχή. Έπρεπε δηλαδή να βρούμε την δυνατότητα να συνδυάσουμε όλες αυτές τις πτυχές, οπότε οι προτάσεις οι οποίες ε, έχουν διατυπωθεί προς εσάς, ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, δεν αποβλέπουν στο να σας προσφέρουν ό,τι χρειάζεστε, αλλά να σας δώσουν πληροφορίες για όλους τους τομείς τους οποίους εξετάζουμε βάσει των οποίων μπορείτε να αποφασίσετε. Συζητήσαμε την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι ένα θέμα που θέλουμε όλοι να συζητάμε και τελικά μας ξεφεύγει ε, διότι πρόκειται για πολύ σοβαρά θέματα ασφαλείας και ε, ε, ε όπως είπαμε παραδείγματο χάρη τι ζημίες δημιουργηθήκαν από το blackout που είχε συμβεί το ίδιο ισχύει και για το ίντερνετ όλα αυτά τα θέματα είναι αποδεχμένα τώρα μέσα για το επίπεδο διαβίωσης το οποίο έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τι πρέπει να γίνει αμέσως τι πρέπει να γίνει στα επόμενα 5-10 χρόνια και ποιο θα είναι ένας πιο μακροπρόθεσμος στόχος που θα μπορέσει να επιτευχθεί σε 15-20 χρόνια. Και βλέπουμε σε όλους τους 95 τομείς ε, ποιες είναι οι προτεραιότητες οι οποίες δεν καθορίζονται μόνο βάσει της βιομηχανίας ε, και της ε, βιομηχανίας ασφαλείας αλλά από ερευνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διάφορους θεσμού με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί για να υπάρχει μία συνέργεια και να επιτύχουμε τις απαντήσεις τις οποίες επιζητούμε. Βεβαίως, θα θέλαμε ε, η μελλοντική μας η μελλοντική μας δραστηριότητα να ε, κατανεμηθεί καλύτερα αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να φτιάξει τέτοιους ε, οργανώσεις παντού. Πρέπει να συνδυάσουμε τους μικρότερους οργανισμούς με μεγαλύτερους και να μπορέσουμε μέσω του Κοινοβουλίου να καταμνήμουμε καλύτερα τους πόρους και ε, ε, ε, τα οικονομικά για να πετύχουμε το στόχο μας. Να εστιαστούμε σε συγκεκριμένες περιοχές, πράγμα το οποίο δεν έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα σημείο εκκινήσεως που δείχνει πώς μπορούμε να κατανείμουμε καλύτερα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως τους πόρους ε, στον τομέα της ερεύνης στο μέλος και βάσει των δύσκολων συζητήσεων που είχαμε καθ' όλη αυτή την περίοδο καταλήξαμε ή στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και να επικεντρώσουμε την ε, ε, χρηματοδότησή μας στην προστασία του πληθυσμού ε, αλλά χωρίς με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε την ακαιρεότητα που επιζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει δηλαδή να ξεπεράσουμε αυτό το όριο ποτέ. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει πλέον να μιλάμε για μια ισορροπία μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ασφαλείας αλλά να πούμε ότι τεχνολογικές λύσεις θα πρέπει να ισχύσουν για μια κατάσταση όπου οι προδιαγραφές που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα παρεμποδιστούν από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνουμε την κατάσταση ε, και εάν δούμε ποιες ε, εταιρείες έπαιξαν σημαντικές κοινωνικό ρόλο θα δούμε ότι όλοι ήμασταν ισότιμοι. Δεν ε, υπάρχει μία πρόταση η οποία ήρθε είτε από μία τεράστια πολυεθνική ή από μία, ένα πολύ μικρό Ινστιτούτο Έρευνας. Προσπαθήσαμε καθ' όλη τη διαδικασία η οποία καθόλου την τη διαδικασια η οποια καταγραφεται στην έκθεση να βασιστούμε σε σωστά επιχειρήματα και ε, στην αρχή της, ε, ε, της συμπεριλήψεως και των τριών πλευρών του τριγώνου στα θέματα έρευνας που μας έχουν απασχολήσει. Οπότε, επαναλαμβάνω, εσείς η πολιτική η αυτή της βάσεως θα μπορέσετε να πάρετε ε, πολιτική απόφαση για να δείτε πού θα διοχετεύσετε τα χρήματά μας, δηλαδή τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Ε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα χωρίς να με έχετε ρωτήσει συγκεκριμένα επ' αυτού. Έχουν υπάρξει προσφάτως πολλές συζητήσεις και μία από τις ερωτήσεις ε, αναφέρθηκε έμεσα μέσα αυτήν την συζήτηση. Δηλαδή, εάν ε, ο τομέας της άμυνας θα χρηματοδοτηθεί περισσότερο, αλλά θα συμβεί ε, το αντίθετο. Εμείς ε, πρέπει να έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση για την προστασία των πολιτών, η τρομοκρατία και η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν είναι τα μοναδικά θέματα που έχουμε να λύσουμε. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και ε, πρέπει να έχουμε τεχνολογίες διπλής χρήσεως, δηλαδή που μπορούν να εφαρμοστούν και σε θέματα ασφαλείας και αμήνης και μιλώντας για το 8ο πρόγραμμα, πλαίσιο πρέπει να εντάξουμε ε, αυτά τα θέματα λίγο περισσότερο στις συλλογισμούς μας διότι αν ε, ε, ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλύτερη χρήση των πόρων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια στην Νότιο Ιταλία είχαμε πάρα πολλά ελικόπτερα τα οποία χρησιμοποιούνται για να κατασβέσουν τις πυρκαγιές αλλά οι πιλότοι των ελικοπτέρων δεν είχαν εκπαιδευτεί ε, για να σβήνουν πυρκαγιές και η επικοινωνία μεταξύ των, ε, ε, ε, των πληρωμάτων των ελικοπτέρων με τις δυνάμεις στην ξηρά δεν λειτουργούσε καλά. Είχαμε, στείλαμε δύο τέτοια ελικόπτερα στην Ελλάδα. Και τι έγινε, μείνανε καθυλωμένα στο αεροδρόμιο επί δύο εβδομάδες λόγω του ότι δεν υπήρχε επικοινωνία. Έτσι δεν μπορείτε να δουλέψετε. Λοιπόν, χρειάζεστε δυνατότητες για να μπορούμε όλοι στις ε, κρίσιμες στιγμές στην καθημερινή ζωή, όχι μόνο σε πυρκαγιές αλλά και σε σεισμούς και σε άλλες φυσικές καταστροφές που διαπιστώσαμε στην Ευρώπη. Ε, σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε ε, εξοπλισμό που θα επιτρέπει την καλή επικοινωνία. Και αυτό είναι το βασικό σημείο το οποίο πρέπει να χρηματοδοτήσουμε στο μέλλον και γι' αυτό θα σας ζητούσαμε να επηρεάσουμε Βάσετε τους ε, υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων για να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση, διότι οι περισσότερες ε, ε, στρατιωτικές εκδηλώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν ουσιαστικά στρατιωτικές επιχειρήσεις, είναι πολιτικές επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγονται από στρατιωτικούς. Δεν έχουμε δηλαδή αρκετό προσωπικό πολιτικής προστασίας το οποίο θα μπορούσαμε να στείλουμε διότι χρειαζόμαστε και κάποιο απόθεμα ε, ε, στην περιοχή μας σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο ατύχημα. Άρα η ανάπτυξη, η βιομηχανική και η έρευνα πρέπει να εξετάσουν και αυτά τα θέματα. Δεν πρέπει να υπάρχουν πλέον κατακαιρματισμοί της βιομηχανίας η οποία ε, συγκρούεται μεταξύ των μεμονωμένων χωρών. Είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουμε. Ότι αντιθέτως οι Αμερικανοί συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και συντονίζουν τη βιομηχανία τους. Οπότε και εμείς θα πρέπει να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να αντιπαραταχθούμε στους εκτός Ευρώπης. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να γίνουν βάσει της αρχής ότι ο τρόπος ζωής μας και οι αρχές μας δεν πρέπει να θυγούν. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο και στον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι ορισμένα ερωτήματα απευθύνθηκαν και σε αυτόν και το δίνω τον λόγο να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια στοιχεία σχετικά με τη φύση του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, Κυρίω για όσου δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Πρόκειται για ένα, έρευνα, ε, για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει οργανωθεί επί τη βάση της πρόκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο, υποβολή προτάσεων δηλαδή, τι οποίε υποβάλλουν ε, εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι με βάση τις δικές τους ε, προτεραιότητες προ την έρευνα, που υπάγεται βέβαια που εντάσσεται μέσα στο πολιτέ πρόγραμμα και που ε, συνάδει με τις προτεραιότητες που έχει ήδη προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από δραστηριότητες όπως αυτές του ΕΣΡΙΦ. Δηλαδή υπάρχουν σαφείς ε, προτεραιότητες Επιτροπής και οι προποθέσει που ορίζει και ο χρήστης, που αφορούν το χρήστη καλύτερα. Και αυτές αποτελούν ε, σημείο εκκίνησης. Το πρόγραμμα πλαίσιο Λέτε, έχει ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Το όντι έχει τέτοια φήμη και σε ορισμένα του σημεία έχει παρεπιστημιακή, δηλαδή ερευνητική περισσότερο κλίση. Ε, αλλά περισσότερο εξαρτάται από τη φύση των, ε, ε, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Και εκεί ακριβώς προσπαθούμε να δώσουμε την έμφαση για να προχωρήσουμε με επιτυχία. Διευκολύνουμε δε την ε, διάδοση των πορισμάτων της έρευνας, που στην τελευταία θα πρέπει να πω δεν είναι και καθήκον της Επιτροπής, είναι καθήκον είτε του δημόσιου τομέα, είτε γενικά των αρχών στην Ευρώπη, εθνικών ή άλλων, αλλά πάντως όχι της Επιτροπής. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε εμείς τη διάδοση αυτών των πορισμάτων με την εμπλοκή του τελικού χρήστη, όπου μπορούμε να τον ε, εντοπίσουμε. Ε, του τελικού εκείνου χρήστη που επί παραδείγματι έχει σαν καθήκον να σώσει ανθρώπινες ζωές, να, να βελτιώσει το επίπεδο της ασφάλειας. Υπάρχουν σαφείς ε, ενδείξεις ε, και προγράμματα που προσελκύουν ασφαλώ τον τελικό χρήστη και μας επιτρέπουν με τον τρόπο αυτό να έχουμε καλύτερα και περισσότερα αποτελέσματα. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή έναν αγαστό κύκλο αντί για ένα φαύλο κύκλο. Ε, προσπαθούμε αυτό να το εντοπίσουμε δε το τελικό χρήστη σε επίπεδο μεγαλύτερων είτε μικρότερων επιχειρήσεων βιομηχανικών. Η, ξέρετε ότι τα θέματα της ασφάλειας έχουν το πολύ πολύ διάρκεια ζωής ε, τριών ετών. Υπάρχει ένα ενδεικτικό όριο για το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε ακριβώς τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου. και θα ήθελα στη συνέχεια να δώσω κάποιες απαντήσεις ως προς την εφαρμογή των ε, πορισμάτων ε, και τι κάνει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω, πρόκειται για αποτελέσματα έρευνας. Η έρευνα αυτή, τα πορίσματα αυτά της έρευνας ανήκουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν υπάρχει ζήτημα πολιτικής, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα ε, ασφάλειας, αλλά ένα πρόγραμμα μόνο ερευνητικό, Όποιο έχει την αρμοδιότητα για την ασφάλεια, οι σχετικέ γενικέ διευθύνσει ή τα κράτη-μέλη με τι αρχέ του, ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την έρευνα. Αυτοί καλούνται να κάνουν τη χρήση τη ε, έρευνα και αντίστοιχα βέβαια σεβόμενοι και τα ζητήματα τα δεοντολογικά ή της ε, του προσωπικού βίου. ως προς την εξωτερική διάσταση της έρευνας ε, και τη διοντολογική είμαστε θυμμένοι να ακολουθήσουμε τις συστάσεις του ΕΣΤΡΙΦ να ενισχύσουμε αυτές τις δύο διαστάσεις στην έρευνα και επίσης θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να διορθώσω τον κύριο Έλλορ για το όσο είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πρόταση για μια προπαρασκευαστική πράξη έρευνα για την ασφάλεια. Το όντι έχει κατευθεί κάπου αυτή η πρόταση. Υπάρχουν πολλέ φήμε που κυκλοφορούν, πλην όμω δεν έχει ε, λάβει η Επιτροπή τέτοιου είδους απόφαση, δεν έχει καταθέσει η Επιτροπή τέτοιου είδους πρόταση. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάτε, θέλετε να επανέλθετε νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και πολύ σύντομα, με μια φράση μόνο. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία δεν θα παραχωθεί σε κάποιο σιρτάρι, δεν θα ξεχαστεί. Έχει αξιοποιηθεί και στο πρόγραμμα Στοκχόλμη και στο ζήτημα του προγράμματος των τηλεπικοινωνιών, της ελληνική διεύθυνση ε, των Επιχειρήσεων ε, και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει ε, εδώ έξω το πλήρες πρόγραμμα που άλλωστε είναι και στη θέση μα του διαδικτύου ή αν θέλετε αφήστε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση να σας το αποστείλουμε. Ή αν θέλετε το δώσουμε στην Επιτροπή και από αυτή να πάρετε τα στοιχεία που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και πάνω απ' όλα για την ε, τροφή για σκέψη που μας προσφέρετε. Ε, μας επισημάνατε ορισμένα ζητήματα. Έχουμε δουλειά και εμείς από πλευρά μας, πράγματα να λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και προχωρούμε στο επόμενο θέμα αμέσως. Ευχαριστώ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διάταξης και θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Μάρτιν Σχούρμαν, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Καινοτομίας και Τεχνολογίας την ΕΙΤΕ, ο οποίος ε, είχε έρθει ήδη να μας δει, έκτοτε όμως έχει εξελιχθεί το Ινστιτούτο του και θα θέλαμε να ενημερωθούμε και θα να δώσουμε την δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής που ενδιαφέρουν για αυτό το θέμα να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους, τον κύριο Σόρμανς που ήρθε εδώ και να του δώσω το λόγο. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη χαρά και τιμή που μου κάνετε μεγάλη την ευκαιρία να συμμετάσχω και πάλι στη συνεδρίασή σας αν μου επιτρέπετε με την πρώτη μου διαφάνεια, να επανέλθω στη βασική ιδέα για το EIT και τα όσα έχουμε προσπαθήσει να επιτύχουμε. Ή τα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Θα σα παρουσιάσω επίση μια επισκόπηση ζητημάτων στο οποίο σα θέλετε να κάνουμε πιστρό διάλογο. Δεν θα μακρηγορήσω, ίσω ε, να περιοριστώ σε 20 μόνο λεπτά για να αφήσω πιστρό χρόνο για τη συζήτηση στη συνέχεια, γιατί είναι πιο σημαντική συζήτηση πιστεύω από την παρουσίαση. Α προχωρήσουμε λοιπόν. Το πιο σημαντικό στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει να δώσω έμφαση πιστεύω, όπως άλλωστε έχουμε δει και στο παρελθόν, είναι ότι η δουλειά μα, η δουλειά του EIT, ως Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι ότι ασχολούμαστε με το τρίγωνο της γνώσης ως ένα σύνολο. Αυτό το υπογραμμίζω για άλλη μια φορά. Γιατί λοιπόν ε, έχουμε επιλέξει την προσέγγιση του τριγώνου της γνώσης, διότι απλούστατα έχει όλα τα στοιχεία αυτό και μόνο αυτό που μπορούν να οδηγήσουν και στην καινοτομία και στην δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα μεγάλα κονδύλια, ούτε τα προγράμματα. Πάνω από όλα εμάς το EIT μας ενδιαφέρει να δημιουργούμε νέα πράγματα, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, νέες, νέα παραγωγή. Ε, κοιτάμε λοιπόν το σύνολο περισσότερο και γι' αυτό θα ήθελα και να υπογραμμίσω ότι αυτό είναι και αυτή είναι η συνδετική ύλη του τριγώνου μας. Και ίσως αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε πάνω απ' όλα, γιατί νομίζω ότι δεν λαμβάνεται αρκετά ε, σοβαρά υπόψη την επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι η συνδετική ύλη. Έχει να κάνει και με την ε, χρήση των αποτελεσμάτων της δηλαδή την, αποτελεσμα... την αποτελεσματική τους αξιοποίηση, αλλά και αποτελεί τον οδηγό που μας καθοδηγεί στην ερευνητική μας δραστηριότητα. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Ε, εφαρμογή λοιπόν των ε, δραστηριοτήτων μας μέσω της ε, καινοτομία και των σχετικών δραστηριοτήτων. Εάν δούμε τις επιδόσεις Ευρώπης ως προς την καινοτομία, και δεν θέλω να επανέλθω στα παραδείγματα που είχα παρουσιάσει και την προηγούμενη φορά, το ότι διαπιστώνουμε ότι έχουμε υστέρηση σε σχέση με τους στόχους που δεν έχουμε ακόμη υλοποιηθεί, πρέπει να εξασφαλίσουμε περισσότερη ε, περισσότερες ικανότητες στην Ευρώπη. Είχαμε μιλήσει με τη Λισαβόνα για το 3% επί του ΑΕΠ που δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε. Είχε γίνει λόγος για το κατά πόσον ήταν σόφρονη η επιλογή του 3%. Εγώ Ω πρόεδρος του EIT, το μόνο που σα πω είναι τουλάχιστον να διατηρήσουμε αυτό και να φτάσουμε στο 3%. Μου αρκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη όμως δεν αρκεί γενικά για τη δουλειά μα το ποσοστό μόνο του 3%. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο εδώ, το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω, ότι δηλαδή πρέπει να είναι ολοκληρωμένο ενοποιημένο αυτό το σύστημα της γνώσης, αυτό το τρίγωνο της γλώσσης. Θα μου πείτε γιατί η εκπαίδευση, η γνώση δηλαδή, να πάει να συνδεθεί με την έρευνα και αυτή ε, επίσης με την ε, επιχειρηματικότητα. Να σας πω. Δεν αρκεί μόνο η καινοτομία ως ε, κρίκος μιας αλυσίδας. Το σύνθημα το οποίο διαρκώς επαναλαμβάνουμε ότι η γνώση, η επιστήμη οδηγεί στην καινοτομία είτε μας αρέσει όχι, ο καθένας με τα γούστα του, έχει χάσει την αξιοπιστία του. Η καινοτομία δεν είναι μόνο επιστήμη και τεχνολογία. Επομένως, χρειάζεται και η διάσταση αυτή βεβαίως, που είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει όμως και η άλλη πτυχή, στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ, με κάπως πιο απερίφραστο, μου επιτρέπετε, τρόπο. Καινοτομία σημαίνει ταυτόχρονα και δημιουργία θέσεων ε, επιχειρηματικής δραστηριότητας καλύτερα. και αυτό συνήθως ε, επιδεινώνεται κατευθείαν αναλογία του αριθμού των, επιχει... των ε, επιτροπών, των συζητήσεων και των κέντρων διαλόγου που αναπτύσσονται. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται ηγετική μορφή, ηγεσία και καθοδήγηση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς με, τις με την κοινότητα των επιστημόνων και μέσα από τα προγράμματά μας. Η ενοποίηση λοιπόν του τριγώνου της ε, γνώσης σημαίνει και καινοτομία, νέα πρότυπα καινοτομία που ενδεχομένω να αποτελέσουν πηγή έμπνευση και για κάποιου άλλου. Και επίση, όπω είπα και στην αρχή, ξέρετε, πολλοί θεωρούν ότι καταρχάς η επιστήμη είναι αυτή η οποία αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της κοινοτομία. Ωστόσο υπάρχει και το κόστος, υπάρχει και η χρησιμότητα, υπάρχει και η πρακτικότητα, υπάρχει και η καινοτομία η οποία γεννάται, κοιτάξτε το παράδειγμα της Κίνας, από την αντιγραφή της καινοτομία των άλλων. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, όλους αυτούς τους παραγόντους πρέπει να τα δούμε. Η καινοτομία λοιπόν ναι, αλλά και η επιχειρηματικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και για να είμαστε ειλικρινεί, κυρίε και κύριοι, στην κοινωνία μα αυτή την εποχή, κοιτάμε τον επιστήμονα, κοιτάμε τον μηχανικό. Εγώ υπήρξα και επιστήμον και μηχανικό. Θαυμάζουμε όμω τον επιστήμονα. Τον επιχειρηματία τον θαυμάζουμε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το μεταστρέψουμε, αυτή την τάση να τη μεταστρέψουμε και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και η επιχειρηματικότητα μέσα στην ε, ανώτατη εκπαίδευση. Τι σημαίνουν λοιπόν αυτές ε, οι ε, η ενσωμάτωση της καινοτομίας σε, στην, τον έλεγχο μάλλον του, τριγώνου της γνώσης σημαίνει να έχουμε εταίρους, εταιρικές σχέσεις αυτόνομες, υψηλής ολοκλήρωσης, με δημιουργικότητα και με διεθνή κατανομή σε θεματικά συγκλίνοντες εταίρους. Αυτό σημαίνει όχι βέβαια εύκολο έργο, την εξέβριση των κατάλληλων εταίρων και μια πολύ σημαντική έννοια την οποία έχουμε εισαγάγει και που επίσης έχει υποστεί αρκετέ επικρίσεις είναι η έννοια της συντοπιότητας ή του συντοπισμού. Αυτό σημαίνει για μένα ότι τα κύρια σημεία του δικτύου της ε, καινοτομίας συνδέονται μέσα από ένα κέντρο, έτσι ώστε η γνώση να είναι δυνατόν να προχωρεί προς την καινοτομία μαζί με τους ανθρώπους που αποτελούν τους φορείς της. Δεν χρειάζονται δηλαδή μεγάλες εκθέσεις, ε, συζητήσεις για μεταφορά κτλ. Όχι, αυτόματα οι άνθρωποι μεταφέρουν τη γνώση. Άλλωστε αυτό δεν είναι και εύρημα της Ευρώπης, δεν είναι εφεύρεση ευρωπαϊκή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ομολογήσουμε, όπως και κάποιες άλλες χώρες, είναι πρωτοπόρες στον τομέα αυτό. Μας έχουν προλάβει και εδώ και αρκετά χρόνια έχουν αναπτύξει αυτές τις έννοιες. Αλλά είναι δύσκολο για μας. Είναι και μεγάλη πρόκληση. Ποιες είναι οι βασικές έννοιες. Μίλησα για την ε, ηγεσία καταρχάς, την ηγετική ε, μορφή ή λειτουργία που αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για μας. Αυτό σημαίνει 20 εταίροι από τους οποίους, στους οποίους καθοδηγεί ένας διευθύνων σύμβουλος και τους ανοίγει το δρόμο, τους δείχνει προς τα που πρέπει να πάνε. Επίσης χρειάζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο όχι ένα πρόγραμμα, αλλά κάτι το οποίο μας δείχνει τι είδους επιπτώσεις θα φέρει η δουλειά που κάνουμε και εστίαση πραγματικά στην, στο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει όχι πόσα θα δαπανίσουμε ή πόσα χρήματα χρειαζόμαστε, αλλά τι θα κερδίσουμε, τι αποτέλεσμα θα μας δώσει. Κοιτάμε λοιπόν το στόχο και πρέπει να είμαστε μερικά χρόνια έτοιμοι να δώσουμε τις απαντήσεις. Μίλησα για την επιχειρηματική δραστηριότητα, το είπαμε, έχει κεντρική σημασία. Επίσης και για το Κοινοβούλιο θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δηλαδή δεν θέλουμε να μας λένε ναι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, αυτό δεν γίνεται, κάντε το διαφορετικά να το συστήσουμε πρώτα. Όχι, εμείς δεν καθόμαστε να κάνουμε τι κουβέντε. Κάνουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε και εσεί μα κρίνετε εκ του αποτελέσματο. Αυτό νομίζω είναι και η βασική έννοια εδώ. Και επίση θέλουμε τα πράγματα να είναι απλά. Εννέα σελίδε η έκθεσή μα, τίποτε παραπάνω. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και επίση σημαίνει ότι παίρνουμε, δεν τρέχουμε κάποιο κίνδυνο, λαμβάνουμε μάλλον κάποιον κίνδυνο, αλλά, είμαστε, αλλά είναι ελεγχόμενο ο κίνδυνο. Τρία θέματα έχουμε επιλέξει στις εταιρικές μας ε, σχέσεις, το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή, την ε, καινοτόμο ενέργεια και τα εργαστήρια ε, πληροφορίας και επικοινωνίας. Τρία βασικά θέματα λοιπόν που έχουμε επιλέξει από το Δεκέμβριο με, τους καθοριστικό παράγοντα, ένα πολύ απλό παράγοντα στην επιλογή από το Συμβούλιο μας, ότι ήταν η υπεροχή ως προς την επίτευξη των στόχων με βάση αυτό το γνώμονα κάναμε τις επιλογές μας. Και πολύ σύντομα επιτρέψτε μου να επισημάνω τι θα κάνουν αυτοί οι εταίροι. Ως προς την εταιρική σχέση του κλίματος, Climate Kick, θα επικεντρωθούμε σε τέσσερις τομείς. Θα αξιολογήσουμε δηλαδή τις κλιματικές αλλαγές και τους φορείς ή τα, στοιχεία που τις, που τις, καθοδηγούν. Θα συζητηθούν επίσης ε, οι πόλεις ε, χαμηλής παραγωγής άνθρακα, προσαρμογή ε, της διαχείρισης των υδάτων και μηδενική ε, παραγωγή άνθρακα ή εκπομπών άνθρακα. Όλα αυτά με το, με το σύστημα του συντοπισμού θα επανέλθω αργότερα. Λονδίνο, Ζηρίχη, Βερολίνο, Μητροπολιτική χώρα, Ράντστατ και αν δεν γνωρίζετε ποια είναι, είναι Μητροπολιτικός χώρος των κάτω χωρών, το Ράντστατ. Και Επιπλέον, πολύ ενδιαφέρον, έχει εισαχθεί επίσης η έννοια των περιφερειακών κέντρων καινοτομία, όπου θα αναπτύσσεται περαιτέρω επεξεργασία αυτών των ιδεών, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όπως βλέπετε είναι κατανεμημένα αυτά τα κέντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και εδώ έχουμε αυτά τα, τα κέντρα συντοπισμού, όπως είπαμε. Έχουμε τα περιφερειακά κέντρα καινοτομία και στο χάρτη βλέπετε ολόκληρη την προσέγγιση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που καθοδηγεί όλες αυτές τις δραστηριότητες υποστηριζόμενος και από την δέσμευση, η ανάληψη από πλευρά των κέντρων συντοπισμού στην επίτευξη σε κάποιους, κάποιων συγκεκριμένων στόχων και ταυτόχρονα και τα περιφερειακά κέντρα καινοτομία τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω αυτούς τους στόχους. Με ένα παράδειγμα, για να μην μακρηγορώ, το οποίο όμως μπορεί να σας δώσει μια εντύπωση. Εδώ έχουμε την, ε, το στόχο της, ε, των ε, προγραμμάτων συστημάτων παραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό το επισημαίνω γιατί έχουμε να κάνουμε μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε εδώ τη Cisco, βλέπετε ονόματα. Πολυεθνική Ευρωπαϊκή Εταιρεία, όπως γνωρίζετε. Βλέπουμε ονόματα όπως η Shell, την Beluga Shipping, βλέπετε την Bayer, την DSMI. DSM μάλλον. Και αυτό που θέλω ακριβώς να σας επισημάνω είναι ότι οι εταίροι που έχουμε επιλέξει και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επιλογή μας έχουν ταυτόχρονα και το χαρακτήρα σημαντικών επιχειρήσεων παραγόντων στον επιχειρηματικό χώρο. Και αυτό είχαμε επισημάνει και από την προηγούμενη φορά. Εφόσον δηλαδή σημαντικές επιχειρήσεις εμπλακούν, θα έχουμε και καλά αποτελέσματα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα και έχει κεντρική σημασία γιατί είναι πολύ σημαντικό η διάσταση βέβαια του επιστημονικού, προσωπικού, του διδακτικού προσωπικού, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε και τους μεγάλους επιχειρησιακούς εταίρους. Ινο, ε, καινοτόμος ενέργεια, Inno Energy. Εδώ πάλι θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ενεργειακό, το οποίο θα επιτρέπει μια ουδέτερη ως προς τις κλιματικές εξελίξεις Ευρώπη μέχρι το 2050. Έχουν προσδιοριστεί τα κέντρα συντοπισμού στην Καλσρούη, την Κρενόμπλ, το Άιτχόφεν, τη Λόβεν, η Λουβέ αν θέλετε, ε, τη Βαρκελόν, την Κρακοβία και τη Στοκχόλμη. Και εδώ ε, συμπληρώναμε μία γραμμή στην διαφάνεια μου ότι ε, ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δραστηριότητε τους με το καταστατικό, με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι του ενδιαφέρει με σοβαρότητα να πάρουν την νομική αυτή μορφή και την οικονομική αυτή, νομική προσωπικότητα και την οικονομική αυτή μορφή. Βλέπετε δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με, με συμπράξει ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχουμε να κάνουμε με πάνω από 20 μεγάλε επιχειρήσει που είναι διατεθειμένε να συνεργαστούν μέσα σε μια νομική προσωπικότητα για να προχωρήσουν στο μέλλον. Είναι μια πολύ, ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, ξέρουμε ότι θα γίνει από την μέρα στην άλλη, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Επίση, ε, κάποια παραδείγματα που μπορώ να σας δώσω για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε Βλέπετε το κέντρο συντοπισμού εδώ κυρίες και κύριοι. Βλέπετε επίσης και την σαφέστατη εμπλοκή των επιχειρήσεων ABP, EDF, SABP της Γερμανίας, η Schneider, μια από τις κύριες επιχειρήσεις. Μεγάλες και ισχυρές επιχειρηματικές ε, μονάδες, επιχειρήσεις. Και δεν τις παρακαλέσαμε. Απλώς εκδήλωσαν μόνες τους το ενδιαφέρον τους, γιατί είδανε ότι υπάρχει ήδη μέσα σε αυτές τις συγκεκριμένες περιφέρειες Ευρώπης η υπεροχή στην καινοτομία και στην έρευνα και στην επιχειρηματική εφαρμογή. Και έτσι τις ενσωμάτωσαν μέσα σε αυτήν την ε, αντίληψη της ε, και της επιχειρηματικότητας. Ε, του EIT δηλαδή. Βλέπετε εδώ η παραδείγματι στην ε, Σουηδία την πρόθεση για ένα FES ηλεκτρικό δίκτυο στην Πολωνία που έχει ήδη αρκετή τεχνογνωσία ως προς τις τεχνολογίες καθαρού άνθρακα. Σας είπα νωρίτερα ότι η Κίνα, στην προηγούμενη μου παρουσίαση εδώ, ότι η Κίνα είναι ο πρωτοπόρος στον καθαρό άνθρακα, ε, αλλά και η Πολωνία έχει πάρα πολύ καλή θέση. Τα ICT Labs, τα, εργαστήρια, τα εργαστήρια πληροφορίες και επικοινωνίας, που επίσης έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί να αλλάξουν και το τοπίο ολόκληρο της Ευρώπης, εξετάζουν την ε, καινοτομία και τον συνδυασμό της καινοτομίας με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που θα οδηγήσει, ελπίζουμε, εφόσον προχωρήσουν και επιχειρήσει όπως θα θέλαμε, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο αυτών των ε, υπηρεσιών που θα είναι στηριγμένε ε, στην διάδοση των, στο, που, ε, θα στηρίζονται στο ίντερνετ. Έχουμε κέντρα στοπισμού, το Βερολίνο, το Άιτχόφεν, το, το Ελσίνκι, το Παρίσι και τη Στοκχόλμη και πάλι έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, τη France Telecom, την Τεχνόπολη, την Κίστα, την Siemens και άλλες που θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν με πιο επιθετικό τρόπο στην καινοτομία στον χώρο της πληροφορίας και της επικοινωνίας, που δυστυχώς κυρίες και κύριοι, ε, δυστυχώς πρέπει να το ομολογήσουμε, ε, στην Ευρώπη έχει, προχωρήσει, έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια εκτό Ευρώπη. Ένα παράδειγμα είναι το Google, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Τέλο πάντων, τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να ξαναδράξουμε την υπόθεση αυτή και να μπούμε μέσα στο παιχνίδι, όπω λέμε. Βλέπετε τα, ισχυρού εταίρου που συμμετέχουν εδώ, Αλκατελουσάν στη Γαλλία, τη Γερμανία, SAP, Siemens. Είμαι ε, βέβαιος ότι θα είναι επιτυχής και αυτή η εταιρική σχέση, αυτή η ΚΙΚ, που έχει επίσης ταυτόχρονα και κέντρα στις άλλες χώρες, σε άλλες χώρες, με στόχο τη διάδοση των ε, πορισμάτων και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει κλάστερ και στην ε, Βουδαπέστη και στην Ιταλία και αλλού. Ε, μια διαφάνεια για το τρίγωνο της γνώσης για μια φορά, για να έχετε μια γενικότερη εικόνα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τη ΔΑΚΙΚΣ, με τις εταιρικές αυτές σχέσεις, είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε νέες μορφές εκπαίδευσης και νέα φουρνιά επιχειρηματιών, νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ευρώπη. Τα πολλά από τα πανεπιστήμια μέσα από τα ΚΙΚ μας έχουν την ίδια αντίληψη ευτυχώ. Είμαστε τυχεροί διότι δεν επιθετική εντό αγωγικών προσέγγιση, ε, αναπτύσσουν δηλαδή επαφέ ε, μέσα από τι σχολέ του για την ανάπτυξη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα στεφτεί με επιτυχία και επίση βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολυτομεακά θέματα τα οποία θα μπορέσουν σε χρόνο να καταλήξουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Και πιστεύουμε ότι με αυτό το τρίγωνο φτάνει τελικά η κοινοτομία στην αγορά. Επίσης στην εικόνα αυτή έχουμε, έχουμε συμπεριλάβει και τους κύριους δείκτες επιδόσεων, τους πτυχιούχους, τα δακτορικά, αλλά πάνω απ' όλα την αξία που δημιουργούν τα ε, σχέδια αυτά, με τις νέες ιδέες και με τις πρακτικές εφαρμογές. Αυτά έχουμε σήμερα, τα τρία κίξ, τα, τις τρεις εταιρικές σχέσεις, τις τρεις κοινότητες γνώσης και κοινοτομίας. Τις βοηθούμε δίνοντάς τους ε, μια ε, υποτροφία εκκίνησης θα λέγαμε, που ξεκινήσανε μάλιστα σήμερα πρέπει να σας πω κυρίε και κύριοι ότι δεν είναι τυχαία αυτή η δουλειά. Ε, έχουμε να κάνουμε πολλούς, ε, πολλούς ε, εταίρους, έχουμε να κάνουμε με τρεις διαφορετικές κοινότητες γνώσης και καινοτομίας. Έχουμε δύο εβδομάδες καθυστέρηση, ίσως κάποιοι να πούνε ότι Κακό είναι που έχουμε δύο εβδομάδε καθυστέρηση, αλλά έχουμε μόνο δύο εβδομάδε καθυστέρηση και νομίζω ότι, αξίζουμε συγχαρητηρίων γι' αυτό, γιατί μιλάμε για τεράστια δουλειά που έχουμε καταφέρει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα προχωρούμε στο επόμενο στάδιο και θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία. Ότι ξεκινάμε τώρα τον Ιούνιο με τις εταιρικέ αυτές, ε, με τις κοινότητες ε, γνώσης και κοινοτομίας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε και την συμφωνία πλαίσιο για, τα, ε, για την επόμενη 7 ετία τον Ιούνιο του 2010 με την Βαρκελόνη και τη Μεγάλη Σύνοδο που θα κάνουμε εκεί θα εορτάσουμε και την, πρώτη, και, την εκκίνησή του, αλλά και την, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα πρώτα διδάγματα της λειτουργίας αυτών των ε, κοινοτήτων ε, που είναι πολύτιμα φυσικά, γιατί ναι, είχαμε επιτυχία ω προ την σύσταση και την ανάπτυξη του δραστηριού του ταχύτατα, αλλά τώρα πια πρέπει να δούμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο γρήγορο, κάτι με πιο αποτελεσματικότητα και μπορούμε να τι βοηθήσουμε αυτέ τι κοινότητε να προχωρήσουν πιο ικανοποιητικά. Αυτά θα μας απασχολήσουν στο καλοκαίρι του 2010. Θα συνεχίσουμε στην παγίωση και την αποκομιδή των διδαγμάτων από τις ε, κοινότητε τη τεχνολογία και τη κοινοτομίας, της και της κοινοτομίας. Ε, ξεκινάμε με την, ε, στα, σε ένα επόμενο βήμα έχουμε και τα, την, τα εγγένεια των γραφείων μας στη Βουδαπέστη. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τις προσλήψεις του προσωπικού μας. Τώρα έχουμε 9 μόνο, θα φτάσουμε στα τέλη του 2010 στους 35 και μέχρι το τέλος του 2011 στους 52 συνεργάτες και ε, προσβλέπουμε σε μια οικονομική αυτονομία ε, αυτό αποτελεί δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να σας πω με ικανοποίηση, όχι μόνο δική μας. Ε, έχουμε ως υποστήριξη, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε, πράγμα το οποίο μας βοηθάει ιδιαίτερα γιατί είναι απαραίτητη για μας η οικονομική αυτονομία και ε, πολύ χρήσιμη για τη δουλειά μας και για τις κοινότητες της γνώσης και της καινοτομία. Σαν πρώτα διδάγματα, τι θα μπορούσαμε να επισημάνουμε. Δεν θέλω να σας πω ότι αυτό το προσεχές εξάμεινο, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 2010, θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις για ε, την ατζέντα τη στρατηγική καινοτομία που θα παρουσιαστεί ταυτόχρονα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία ε, με την προοπτική ε, της κοινωνία πληροφορίας. Πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να αντιληφθείτε ότι ο επόμενο γύρο χρηματοδότηση πιθανών τέτοιων κοινοτήτων αφορά το 2014 τώρα. Αυτό που σχεδιάζουμε τώρα αφορά το 2014. Την προηγούμενη εβδομάδα έλαβα δύο προτάσεις για κοινότητες γνώσης και κοινοτομίας που θα ήθελα να ξεκινήσουν τώρα. Εμείς ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε συχνά ε, τηλεφωνήματα από κάποιου που μα λένε: Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδέα να, να έρθουμε να σα μιλήσουμε, να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι για το 2014. Άρα, ζήτημα για μας είναι να καλύψουμε το χρονικό αυτό διάστημα. Το καλό βέβαια είναι ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια μας δίνουν το χρόνο και να ε, διδαχθούμε, να, συγκεντρώσουμε εμπειρία. Ταυτόχρονα βεβαίως κοιτάμε, αναζητούμε και ευκαιρίες να διατηρήσουμε αυτή την ορμή που χαρακτηρίζει τη διαδικασία σε αυτό το στάδιο, ε, ίσως με την... Ε, με μια φάση κυοφορίας θα έλεγα μέσα στο 2012, 2013 έτσι σιγά σιγά να προετοιμαστούν όλα αυτά για να βγουν στην ε, πρακτική εφαρμογή το 2014, στην, στην ουσία δηλαδή το 2014. Όλα αυτά τα δούμε, ε, έχουμε και τη χρηματοδότηση φυσικά ως ζήτημα και όλα αυτά. Πάντως υπάρχουν ζητήματα ε, τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε στο χρονικό αυτό διάστημα. Έχουμε επίσης για το πρώτο ήμιση του 2011 τη διάσκεψη των εμπλεκομένων για την ατζέντα, στρατηγική ατζέντα καινοτομία, το SIA δηλαδή, με την Επιτροπή, με το Κοινοβούλιο, που θα υποβάλει μετά τι προτάσει του Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και επίση θα ήθελα να πω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά πλέον. Στην, είναι, έχει μακρά πορεία του πλέον πίσω το ίδρυμα του IT. Μέχρι το καλοκαίρι πιστεύω θα έχουμε ε, ένα πρόσθετο μέσο με το ίδρυμα για το EIT που θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και των ε, κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, αλλά και τη συνέχιση των εργασιών του EIT. Ταυτόχρονα όμως αυτό θα απαιτήσει και περισσότερα χρόνια, διότι θα πρέπει να χαλιβδώσουμε το, το Ίδρυμα, να εξασφαλίσουμε την ε, προστασία του και την ε, απρόσκοπτη λειτουργία του. Αυτά είχα να πω προς το παρόν επισημαίνω ότι μαθαίνουμε ακόμα τι έχουμε να κάνουμε. Ευτυχώς ε, έχουμε ως στόχο όχι τόσο το πρόγραμμα όσο το να καθοδηγήσουμε τις εργασίες μας προς κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ, ελπίζοντας ότι θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σούρμανς, Θα παρακαλέσω να είμαστε λίγο σύντομοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ε, μισή ώρα μέχρι τι 5 μόνο για τις συζήτηση, γιατί μετά έχουμε και κάποιον άλλο ξένο προσκεκλημένο και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ε, χωρίς καθυστέρηση. Βλέπω ότι έχει ήδη φτάσει, καταφτάσει καλύτερα. Έχω περίπου 10 εγγεγραμμένου για τη συζήτηση και θα ήθελα να παρακαλέσω του συναδέλφου να είναι στο δυνατόν πιο ε, συνεκτικοί στις παρατηρήσεις του. Κυρία Καβάλια, καταρχά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σούρμαντ για την ε, παρουσίασή του και για να τον συγχαρώ για το EID και για την ε, ομαλή έναρξή του. Ήταν ένα δύσκολο πρόγραμμα ε, στο ξεκίνημά του, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ιδιαίτερως ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο έχει προχωρήσει η διαδικασία και κυρίως με την ανταπόκριση των ενδιαφερομένων ε, σε αυτή την ε, πρόσκληση. Ε, κατά την άποψή μου ένα βασικό σημείο για την επιτυχία του EIT ήταν το γεγονός ότι ενδιαφέρονταν γι' αυτό καλά πανεπιστήμια και η βιομηχανία και ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση. Πλέον πρέπει να παγιωθεί η λειτουργία των ΚΙΚΣ, να ετοιμάσετε την ατζέντα για την καινοτομία, αλλά κατά, κατά με η αποστολή του EIT πηγαίνει πέρα από αυτό και θα πρέπει να αποτελέσετε καταλήτη για τον εξυγχρονισμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και καταλήτη για τις σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας. Επιπλέον θα πρέπει να συνεισφέρετε στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας ή όπως ε, εσείς πολύ καλύτερα λέτε στον ευρωπαϊκό χώρο καινοτομίας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Πώς θεωρείτε ότι το EIT μπορεί να ε, πληρώσει το στόχο του, το ρόλο του, να συνεισφέρει στον ευρωπαϊκό χώρο καινοτομίας και κατά πόσον διαβλέπετε κάποια πιθανότητα να γίνονται κάποιες κοινέ ή παράλληλες δράσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και μέσω αυτής της συνεισφοράς να ενισχυθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Καινοτομίας. Ευχαριστώ. η Αγγέλικα Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που ήρθατε. και για την ενημέρωση που μας δώσατε για τις ε, εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια πρώτη ερώτηση λοιπόν, η οποία έχει να κάνει με τη συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στα ΚΙΚΣ Πρόκειται σε τελευταία ανάλυση για τους φορείς της καινοτομίας. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν συμμετέχουν και σε ποιο βαθμό, σε ποια κλίμακα και επίσης εάν είναι μόνο χρηματοδότης, εάν είναι δηλαδή ίδρυμα χρηματοδότηση μόνο το ίδρυμα του EIT, αν έχει και άλλες δραστηριότητες για την καινοτομία. Εδώ πολλές φορές γίνεται λόγο στα κράτη-μέλη ως ε, ε, για πρωτοβουλίες cluster. Αυτό είναι αυτό που κάνετε ή είναι κάτι διαφορετικό. Κύριε Σφανής Ρόι. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω στα Ολλανδικά, διότι άλλωστε και ο κύριος Σούρμεντ μπορεί να με καταλάβει. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για τους ε, ρυθμούς σας. Ε, πραγματικά βλέπουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα κυρίως σε σχέση με τα όσα έχετε επενδύσει. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δεν κάνετε σίγουρα αυτά που κάνουν άλλοι, αλλά πραγματικά εργάζεστε ε, πολύ εντατικά σε θέματα που αφορούν στο κλίμα και τις καινοτομίες. Η δημοσιογράφοι ήταν ενθουσιώδης. Διάβασα στο τύπο ότι χρειάστηκε να του σταματήσετε ε, διότι ήθελαν να συμμετάσχουν όλοι σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού που κάνατε. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε κάποια πράγματα όσον αφορά στη χρηματοδότηση. Τι δέσμευση έχει αναλυφθεί και τι αναμένεται. Δυστυχ, ε, τα κονδύλια αλλάζουν από κικ σε κικ. Και τέλος μια ερώτηση για την καινοτομία. Μας ενδιαφέρει η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η προσέγγιση που ακολουθείτε. Η συγκέντρωση βοηθά για να δημιουργηθεί η κατάλληλη μάζα, κρίσιμη μάζα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουμε εξαιρετικό know-how, αλλά το να μεταλαμπαδεύσουμε κι αλλού ίσως είναι το πιο δύσκολο σημείο της δουλειάς μας. Μπορείτε να δημιουργήσετε συνέργειες με άλλα προγράμματα και σχέδια τα οποία έχουμε υπατμών για το σκοπό αυτό. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές ε, πλατφόρμες. Είναι πράγματα τα οποία είναι αποσυνδεδεμένα ή όλα είναι μαζί στον ίδιο χώρο και γίνεται μια κατανομή αρμοδιοτήτων ε, μεταξύ ημών. Ε, θα ήθελα να ξέρω γενικώ τι θα γίνει γιατί με ενδιαφέρει και για το, μετά το 2013. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ ονόματο τη ομάδα μου να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα για άλλη μια φορά εδώ στην Επιτροπή μα και να σα συγχαρώ για τι εργασίε σα. Ε, Ω συνήθω ε, θα πρέπει να πω ότι συμφωνούμε απολύτω στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε κι εσεί ε, την επιστήμη και την καινοτομία. Μετά από όσα άκουσα λοιπόν και μετά από όσα μα είπατε για τα όσα έχετε κάνει μέχρι τούδε, θα ήθελα να σα ρωτήσω και κατά πόσον θεωρείτε ότι το Ινστιτούτο καλό θα ήταν να ε, βρισκόταν στον αρμόδιο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τη σκέψη της Επιτρόπου Αρμόδιας για την Έρευνα και την Καινοτομία και όχι εκεί που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Επίσης θα ήθελα να σας θέσω δύο επιπλέον ερωτήσεις. Η μία αφορά τη σχέση με την εμπειρία σας για την έναρξη του EIT και ε, με, την, με τις πρώτες προσκλήσεις. Όπως ξέρετε, ε, βρισκόμαστε εν πλήρη συζήτηση για την ε, ε, διαδικασία και την υλοποίηση των όσων έχουν αποφασιστεί στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον κάνατε κάποια πρώτερη εργασία, κάποια πρώτερη ανάλυση για να αποφύγετε το υπερβολικό γραφειοκρατικό ε, για τους εντολοδόχους και επίσης κατά πόσον ελήφθησαν μέτρα ε, τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς στη συζήτηση που κάνουμε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Να, το να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε και να γνωρίζουμε βέλτιστες πρακτικές πάντα είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Μάθαμε ότι απορρίφθηκε κάποιο πρόγραμμα με το επιχείρημα ότι συμμετείχαν και δημόσιοι οργανισμοί σε αυτό. Και γιατί, και σας παραθέτω, θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος πολιτικής επιρροής, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσκομα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή η απάντηση από πλευρά CIT με εξέπληξε, διότι αυτό είναι σε πλήρη αντίφαση με τα όσα έχει ε, δηλώσει το EIT στην προηγούμενη πρόκλησή του που λέει ότι όσοι θα επιλεχθούν σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία καθορισμού των αρμοδιοτήτων και των προτεραιοτήτων συγγνώμη, έρευνας και τεχνολογίας. Όντω ισχύει αυτό ή θα μπορούσατε να μου επαληθεύσετε ότι ισχύει ή να μου το διαψεύσετε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, το Ίδρυμα που εκπροσωπείται ε, αναπτύσσει δραστηριότητα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα της έρευνας και θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, μπορούμε να ενημερωθούμε για την ε, κατάσταση και των πανεπιστημίων στον ερευνητικό χώρο. Μιλήσατε για το τρίγωνο της γνώσης. Μιλάμε συχνά για το επιστημονικό, για το τρίγωνο τη επιστήμη, τουλάχιστον στο έκτακτο πρόγραμμα πλαίσιο. Συγκεκριμένα αποτελέσματα λοιπόν, απτά αποτελέσματα μπορείτε να μας δώσετε για να μας δείξετε, να μας αποδείξετε ότι έχετε επιτύχει κάτι συγκεκριμένο. Όχι γενικές απαντήσεις, αλλά συγκεκριμένες παραμέτρους με τις οποίες να μπορούμε να προσμετρήσουμε τις επιδόσεις αυτών των ερευνητικών κέντρων. Ε, είπατε ότι έχετε επίσης, δεύτερη ερώτηση, εννέα συνεργάτες. Ποιος μπόρεσε να οργανώσει αυτές τις κοινότητες με μόνο εννέα συνεργάτες, πώς τα καταφέρατε. Τρίτη ερώτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, του Προεδρείου. πολύ σημαντική ε, λειτουργία ασφαλώς έχει, πολύ σημαντικό ρόλο. Μάθαμε, ακούσαμε ότι υπήρξε κάποιο ζήτημα πολιτικής επιρροής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχει η περίπτωση να εκπροσωπείται κανείς στο Συμβούλιο, όχι με κάποιο κράτος, όχι με επιστήμονα, αλλά με ε, πολιτικό. Κυρία Τιτσάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σούρμανς ε, για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσε και θα είχα και κάποιες ερωτήσεις. Η μία αναφέρεται στην γεωγραφική συνεργασία ένα θέμα το οποίο ανέφεραν και δύο συνάδελφοι πριν. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν κύριε Σούρμαντς κατά πόσον ε, θεωρείτε ότι είναι σωστό να μην υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη. Για ποιο λόγο δεν έχουμε εκπροσώπους από αυτά τα κράτη-μέλη και γιατί θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι φραγμοί ε, που δεν επιτρέπουν ε, να συμβαίνει κάτι τέτοιο και τι θα θέλετε να, τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση για την... Ε, Διανοητική ιδιοκτησία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο ιδιωτικό τομέα ε, συμμετέχει ενεργά. Είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθεί ο ιδιωτικό τομέα. Αλλά εάν δεν υπάρχει γεωγραφική κάλυψη που να ε, καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε κέντρα ανταγωνιστικότητας ει βάρο άλλων. Παραδείγματο χάρη να έχουμε το χ σε κάποια περιοχή που θα σημαίνει ότι κάποια άλλη περιοχή θα είναι λιγότερο ευνοημένη. Σα ρωτώ λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε με θέματα διανοητικής ιδιοκτησία και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στην Ευρώπη. Κάτι επιπλέον, σας παρακαλώ μην ξεχάσετε να απαντήσετε στην ερώτησή μου γιατί δηλαδή θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορέιρα Τεκάμπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση. Πριν από την ερώτηση όμως, πρέπει να σας πω ότι είναι η δεύτερη φορά που σας ακούω και κάθε φορά χαίρομαι ακόμα περισσότερο που σας ακούω. Επομένως, συγχαρητήρια κύριε Σούρμαντς. Και τώρα η ερώτησή μου. Η ερώτησή μου αφορά αυτό το ηγετικό μοντέλο και την, ε, το διευθύνοντα σύμβουλο, τον CEO. Ο κύριος ε, Σούρμαντς μας είπε ότι έχει τυφλή ε, εμπιστοσύνη στην ηγεσία και λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο. Πώς όμως μπορεί ένας διευθύνοντας σύμβουλας να ηγείται ενός ε, συνόλου οργανισμών που ο καθένας έχει διαφορετικές αρμοδιότητες εάν τα μέσα τα οποία διαθέτει ε, το οπλοστάσεό του δεν είναι παρά ένας ελάχιστος προπολογισμό πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να υπερβείτε το πρόβλημα και ε, να μην ε, έχετε τις δυνατότητες που πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Κύριε Σούρμαντς, εδώ είμαι. Ναι. Ε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εγώ για την παρουσίαση. Είχα και εγώ την ευκαιρία να μελετήσω τις δραστηριότητες του EIT και πρέπει να πω ότι ήταν ε, εξαίρετε οι εντυπώσει που Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. πρώτη ερώτηση που με απασχολεί ήδη καλυφθήκε από του συναδέλφου Έχει να κάνει με τη γεωγραφική πτυχή. Πώς λοιπόν μπορεί το όνσιτο σας, η δουλειά σας ε, να ε, είναι πιο αποτελεσματική ως προς τα ε, κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία ξέρουμε ότι χωλένουν ως προς το τρίγωνο της γνώσης εδώ. Είπατε ότι πρόκειται για τη σχέση μεταξύ της γνώσης και της καινοτομία, που είναι συχνά ε, ελλειπής, όπως επίσης και τη σχέση μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να επιδιώκουμε... Ξούμε να επιδιωχθεί η ομοιογένεια και ε, πρέπει και κάποιος να διαδραματίσει τον ηγετικό ρόλο. Ιδιαίτερα δε, με χαρά, ε, άκουσα ότι σε δύο εβδομάδες, λέει θα ανοίξετε και, και το, θα κάνετε και τα εγγένεια του κέντρου σας ε, στην Βουδαπέστη. Πιστεύω ότι και αυτό θα μπορέσει να προσφέρει στις εργασίες σας ιδιαίτερα. Έχω δε μια ερώτηση Η τεχνολογία ε, χαμηλών εκπομπών ε, άνθρακα, είπατε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος, αλλά ε, υπάρχουν άλλοι. σκοπεύετε παραδείγματι να ασχοληθείτε με τους αντιδραστήρες σύνδεξης, πυρηνικούς αντιδραστήρες σύνδεξης. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να δώσουμε και στον κύριο Σνόρμα τη δυνατότητα να απαντήσει για να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Α, έχετε και εσεί μια ερώτηση ακόμη, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, Ευχαριστώ πολύ. Ελίζα Μπόμεν από την Επιτροπή των Περιφερειών. Και θα ήθελα να ζητήσω και κάποιες ε, πληροφορίες επιπλέον, να μας πείτε κάποια επιπλέον στοιχεία για τα κέντρα καινοτομία. Και τώρα Well, first of all, thank you very much. Ευχαριστώ. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ε, ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις πάρω με τη σειρά. Να ξεκινήσω με τις ε, ερωτήσεις που μου κάνατε για το ERA και το τι θα μπορούσαμε να μάθουμε από την προσέγγιση του EIT. Σαφώς δεν βλέπω κάποιες δυνατότητες και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το εστιάσουμε σε δύο διαφορετικούς τομείς. Το ένα είναι το Συμβούλιο Έρευνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο ε, φέρνει εξαίρετους ε, επιστήμονες από όλη την Ευρώπη και φαντάζομαι ότι τελικώς αυτό θα πρέπει να συγκεραστεί με την καινοτομία. Ε, παρά το γεγονός είπα ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν οδηγεί στην καινοτομία, νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να εξετάσουμε τουλάχιστον κάποια στοιχεία αυτών των προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα Έρευνας και εγώ ε, τίνω να την αποκαλώ ατζέντα έρευνας και όχι καινοτομίας μόνον. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, σαφώ η εκπαίδευση θα πρέπει να περάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Για την επιχειρηματικότητα έχω διαπιστώσει σε πολλέ χώρε ανά τον κόσμο ότι ε, εμείς είμαστε πίσω, ε, πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, κάποια εξαιρετικά πανεπιστήμια στα ΚΙΚΣ τα οποία θα μπορέσουν να αναπτύξουν σημαντικά στοιχεία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τα φέρουμε όλα αυτά στον τομέα της καινοτομίας γιατί είναι θέμα ε, της ε, έρευνας που κάνουμε και η παιδεία, η κατάλληλη παιδεία. Τώρα, για τόσα θέλουμε να κάνουμε για το μέλλον, νομίζω με ρώτησε και η κυρία Νίμπλερ για τη χρηματοδότηση. Πού είναι η κυρία Νίμπλερ? Α, να βλέπω τώρα. Η χρηματοδότηση είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν είναι ασήμαντο. Ε, επιτρέψτε μου να μην σας πω πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Έχουμε σαφώς ε, ιδέες για το πώς ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά βρισκόμαστε στο σχέδιο, των, στη φάση των ιδεών και μόνον αυτή τη στιγμή, όχι στην υλοποίηση. Ελπίζω ότι θα γίνει και θα είναι και αρκετά ισχυρό, ώστε για να έχει και τις κατάλληλες επιπτώσεις. Για τα κλάστερς, το είπα αυτό και πριν από κάποιους μήνες, πραγματικά πιστεύω ότι η πολιτική των clusters είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη. Ειλικρινά το πιστεύω. Βέβαια, οι πολιτικές κλάστερς έχουν και περισσότερες ε, συνέπειες, και εδώ έρχομαι και στην ερώτηση του κυρίου Φανερίστερ Ρόι, όταν μπορούμε ε, να έχουμε και την ιδέα του συντοπισμού. Ε, οι περιοχές οι περιφέρειες τη σήμερα ημέρα έχουν πάρα πολύ την έννοια αυτό του θα συνεργαστούμε και αυτό είναι. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε και τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν μπορεί ένα κλάστερ στην Ευρώπη απλώς να πηγαίνει από με τον τρόπο με τον οποίο συζητάτε τα τελευταία χρόνια και τελικά να μην υπάρχει κάποιος προσανατολισμός για το στόχο. Ε, το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει σημασία κυρίες και κύριοι. Εγώ να πω ότι είμαι υπέρ του αποτελέσματος αλλά θα πρέπει να είμαστε και προσανατολισμένοι προς το αποτέλεσμα. Ο κύριος Φανίστεν Ρόι επίσης με ρώτησε για τι ε, επιπτώσεις του ΦΠΑ. Έχουμε 390 εκατομμύρια ευρώ όπως θα γνωρίζετε όλοι χρηματοδοτούμε μόνο το 25% των δραστηριοτήτων, που σημαίνει το 75% των δραστηριοτήτων είναι δέσμευση των συμβαλωμένων μερών. Και επίσης, ξέρετε ότι θα υπάρξει και χρηματοδότηση από τα διευθυντικά ταμεία και το Ταμείο Έρευνας και Ανάπτυξης, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να συνεισφέρουν αυτοί. Ε, η ιδέα αυτού του τριγνώνου γνώσης, ε, του ηγετικού ρόλου, το η έννοια ότι άλλες χώρες κινούνται πιο γρήγορα από ότι εμάς στην Ευρώπη είναι σημαντικό και πραγματικά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη προθυμία, μεγάλη διάθεση να προχωρήσουμε. Και επίσης πιστεύω κάτι το, ότι κάτι το οποίο άλλαξε ε, τα πράγματα σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν αυτή η έννοια του συντοπισμού μέχρι πρόσφατα, 1,5 περίπου χρόνο νομίζω, στην Ευρώπη ε, λέγαμε ότι πρώτα θα πρέπει να γεννήσουμε τη γνώση και μετά θα πρέπει να βρούμε πού θα πρέπει να δοθεί και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Η ιδέα του συντοπισμού είναι ακριβώς ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούν για το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν ε, προσμετράτε λοιπόν μόνο αυτό που δίνουμε, μετράμε και το αποτέλεσμα και αυτή είναι η βασική έννοια. η προσέγγιση αυτή είναι τελείω διαφορετική. Θα ήθελα να τη συζητήσω κάποια άλλη στιγμή. Είναι μια τελείω διαφορετική προσέγγιση και δεν θα ήθελα να σταθώ εδώ σε αυτό. Αλλά να πω ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία κάνουμε εμεί ε, στο EIT ε, γίνεται και στα κοινά κέντρα ερευνών, στα JTI, αλλά ε, ο δικό του ο ρόλο είναι τελείω διαφορετικό. Εμεί είμαστε πειραματικό οργανισμό, η δική του προσέγγιση διαφέρει. Εκτιμώ το γεγονό ότι ήσασταν τόσο ειλικρινεί ε, και θέσατε αρκετοί από εσά το θέμα της ε, γεωγραφική κάλυψης. Ενδιαφέρον είναι αυτό, αλλά το EIT δεν αφορά τη γεωγραφική κάλυψη. Σα το δηλώνω αυτό ξεκάθαρα. Το EIT θέλει να έχει αποτελέσματα σε τρει τομεί που έχουν επιλεχθεί αυτή τη στιγμή από εσά, ε, κυρίω το κλίμα, την ενέργεια και την, έρευνα, την πληροφορία και τις επικοινωνίες και έχουμε επιλέξει τα ΚΙΚΣ μόνο βάσει της αριστείας που έχει ήδη επιτευχθεί και σε θέματα εταιρικών σχέσεων και σε θέματα καινοτομίας για να επιτύχουμε το στόχο μας. Και αυτό ήταν το κυρίαρχο κριτήριο το μόνο και κυριαρχό κριτήριο ε, ήταν μια πολύ ανοιχτή διαδικασία. Καταλήξαμε σε έξι προτάσεις τελικά τα οποία οι οποίες συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόταση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Μαντουρέλ δεν ήταν μία από τις έξι, είχε απορριφθεί νωρίτερα στη διάρκεια της πρόσκλησης και οι έξι αυτές προτάσεις ε, συζητήθηκαν, έγιναν συνεντεύξεις, έγινε μία σύντομη συζήτηση έγινε μία και μόνη μυστική ψηφοφορία ώστε να μην μπορεί να επηρεάσει κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του άλλου. Δεν υπήρχε κανένας που να μην συμμετείχε στις συνεντεύξεις και στις ε, ε, τελικές διαδικασίες που να έχει συμφέροντα επί του θέματος και τελικά μετά από αυτή τη μία και μοναδική ψηφοφορία αποφασίσαμε. Είναι μία απλή, διάφανη και γρήγορη διαδικασία. Ε, ίσως να καταλήξει κάποιος στο συμπέρασμα ότι ίσως να μην έχουμε την τέλεια γεωγραφική κάλυψη μετά από τα αποτελέσματα που είχαμε. Ε, υπάρχουν όμως ένα-δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω εδώ. Πρώτον, τα kicks δεν θα είναι τα ίδια ε, σε χρονικό ορίζοντα, σαφώς θα υπησέλθουν αλλαγές και αυτό φυσικά θα οδηγήσει και σε νέες συνεισφορές από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης στο μέλλον μία παρατήρηση αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αν τα kicks κάνουν τη δουλειά τους καλά, αυτό θα μας οδηγήσει σε ε, παραδείγματα και γόνιμα ε, στοιχεία ως προς το κόστος για χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή είτε δεν συμμετέχουν καθόλου είτε δεν συμμετέχουν τόσο ενεργά. Ε, να πω ότι η Πολωνία υπάρχει, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία. Δεν θα πρέπει να είμαστε και τόσο αρνητικοί για τη γεωγραφική κάλυψη. Νομίζω ότι είναι αρκετά ευρεία η κάλυψη. Αλλά αν δεχτείτε την έννοια του συντοπισμού, η γεωγραφική κάλυψη ποτέ δεν θα είναι τέλεια. Αν θέλετε να έχετε γεωγραφική κάλυψη, δεν μπορείτε να έχετε συντοπισμό, διότι εκεί χάνετε το σημείο εστίαση και η όλη ιδέα δεν θα λειτουργήσει. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω μια πολύ σαφή απάντηση επί του θέματος και αυτή ήταν η απάντησή μου. Τώρα, για την ηγεσία. Πώς μπορείτε να έχετε τέσσερα ή πέντε διαφορετικά υποθέματα εκεί και σε διαφορετικά κέντρα συντοπισμού. Αυτή νομίζω ήταν η ερώτησή σα. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και με ένα διευθύνοντα σύμβολο μια επιχείρηση, ο οποίο πρέπει να ασχοληθεί με 4-5 διαφορετικά τμήματα. Αυτό ο άνθρωπο θα πρέπει να κρατά μια σχετική απόσταση από τα όσα συμβαίνουν και θα πρέπει να έχει ανθρώπου σε κάθε κέντρο που θα κάνουν τη δουλειά του. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει εμένα δεν είναι τόσο αυτό, όσο το γεγονό ότι θέλουμε να έχουμε κάποιο κόσμο και να διασφαλίσουμε ότι ακόμα και η βιομηχανία τα δεν γνωρίζει αυτή την έννοια της ηγεσία. Και εγώ έχω μιλήσει με μέρη του, της βιομηχανίας όπως και με άλλους ενδιαφερομένους και πάντα η βιομηχανία λέει προτιμούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι σαφώς προσανατελεσμένο στο αποτέλεσμα και θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα αναλάβει τα ενία παρά κάποια προγράμματα στα οποία θα συνεισφέρουμε και εμείς και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Επομένως, Θέλουμε όλοι αποτελέσματα. Και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Μίλησα με όλους τους ε, διευθύνοντες συμβάλλους, τους τρεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και τα πράγματα είναι καλά και νομίζω ότι με χαρά θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι το βασικό εδώ. δεδομένα τα οποία μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε. Νομίζω η ερώτηση ήρθε από εσά, ε, κυρία μου. Δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό. Πώς να το πω ε, με ωραίο τρόπο τώρα. Έχουμε την τάση στην Ευρώπη να εξετάζουμε δραστηριότητες, προγράμματα, έργα και να πηγαίνουμε απευθείας στα στοιχεία που θα προσφέρουμε. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Το να κοιτάει κάποιος τα αποτελέσματα ε, τα επιχειρηματικά αποτελέσματα κλπ. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και αν μιλήσετε με ανθρώπους του ΟΣΑ, διότι το έχουμε κάνει αρκετές φορές πλέον αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια και είναι περίπλοκα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε προετοιμάσει, δεν θα σας τα δώσω τώρα, αλλά έχουμε προετοιμάσει έναν απλό πίνακα αποτελεσμάτων, ώστε τα κίξ μας να μετρούν τα αποτελέσματά τους θα ήθελα σίγουρα να σας το παρουσιάσω αυτό, κύριε Πρόεδρε, στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι τα ΚΙΚΣ έχουν τα δικαιώματα συζητήσεων μαζί μας πρώτα. Θα πρέπει να αποφασίσουν ε, ποια είναι οι βασικοί δείκτες απόδοσης και από εκεί και πέρα θα τους έχουμε στον πίνακα αποτελεσμάτων. Θα έχουμε 4, 5, 6 ενδεικτικά στοιχεία απόδοσης και θα μετρούμε ανελαίητα τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή, η ετήσια επιδότηση θα εξαρτάται και από την απόδοσή τους. Ε, έτσι θα υπάρχει και κάποιος ανταγωνισμός και ε, μπορεί να έχουμε 6-7 κίξ ε, τα οποία θα έχουν κάποιον ανταγωνισμό. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Θα σταματήσω να απαντώ ερωτήσεις γιατί νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζητά να προσθέσει κάτι, οπότε ε, έχουμε ολοκληρώσει ε, όπως ε, είπε και ο κύριος Κάμπας θέλω να ευχαριστήσω διότι δεν είναι μόνο ενδιαφέρον αλλά και ικανοποιητικό να ακούει κανείς όχι μόνο τις καινοτομίες αλλά να αντιλαμβάνεται τις ιδέες και είναι διάφορα θέματα που, στα οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο ε, μετά θα μπορέσει να επαναφέρει την Ευρώπη στο προσκήνιο της καινοτομίας στην Ευρώπη πρέπει να αποβλέπουμε στην αριστεία και στα βέλτιστα αποτελέσματα. Και για να το επιτύχουμε θα χρειαστεί να αναλάβουμε κινδύνους. Στην αρχή ήμουν αρκετά κατακριτικός, αλλά τώρα ακούω ότι ε, όσο περισσότερα ακούω τόσο περισσότερο πιστεύω ότι η μεθοδολογία αυτή μπορεί να μας βοηθήσει για να ενημερωθούμε και για άλλα προγράμματα. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και δέστε τι μπορείτε να κάνετε και για τα άλλα προγράμματα και ίσως μπορούμε να επανέλθουμε στα θέματα αυτά και πάλι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Meine Damen und äh, συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε πάλι, διότι νομίζω τελειώσαν οι φωτογραφίσεις τώρα και θέλω να καλωσορίσω κάποιον εδώ σήμερα τον οποίο δεν βλέπουμε κάθε μέρα είναι ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργείας, ο κύριος Τανάκα ο οποίος στον τομέα της ε, ενεργειακής ανάλυσης και πολιτικής είναι ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο και όλοι όσοι πρόσεξαν κάπως και έχουν διαβάσει γνωρίζουν ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμμετέχει στη χώρα του στο πολιτικό τομέα, στα θέματα του περιβάλλοντος και χαίρομαι πολύ που ήρθε εδώ και λυπούμεθα γιατί ε, χρειάστηκε να σας βάλουμε στο τέλος της ημερησίας διατάξεως. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι του ύψου σας, αλλά δεν θέλαμε να μην σας δούμε καθόλου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ε, κάποια ενημέρωση, οπότε σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας, για το χρόνο σας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας πείτε κάτι καινούριο που να έχει σχέση με τις ε, προοπτικές ε, της ενεργείας του 2009 και ε, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε κάποιο χρόνο να σας ακούσουμε, να μας πείτε ε, τα γεγονότα και τους ε, αριθμούς και μετά να αποφασίσουμε. Δηλαδή να μην αποφασίζουμε πολύ γρήγορα, αυτό είναι λάθος. Οπότε σας ευχαριστώ που ήρθατε και έχετε το λόγο. Δυστυχώς δεν μπορείτε να μεταφράσετε τα Ιαπωνικά. Προσπάθησα να δω εδώ την, τα Ιαπωνικά στη μετάφραση, αλλά δεν είναι ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ιαπωνία, οπότε θα χρειαστεί εγώ να μεταφράσω τον εαυτό μου και σας παρακαλώ να αντέξετε και να υπομείνετε τα κακά μου αγγλικά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Ρόιλ που με καλέσατε να μιλήσω στην Επιτροπή σας ε, για την έρευνα και τη βιομηχανία και την ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ο οργανισμός μας δημιουργήθηκε το 1974 από πολλούς ε, από τους ε, συναδέλφους σας και από όλες τις ε, ανεπτυγμένες χώρες της εποχές, την Ιαπωνία, την, τις Ηνωμένε Πολιτείες, διότι θέλαμε να καταρτήσουμε σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης να έχουμε ένα απόθεμα πετρελαίου 90 ημερών ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε έκτακτες περιστάσεις. Ε, η οργάνωση εδρεύει στο Παρίσι, είναι ε, μία αδελφή οργάνωση του ΟΣΑ και αναφέρεται στην ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε χρησιμοποιήσει δύο φορές στην ιστορία μας αυτό το στρατηγικό απόθεμα. Μία φορά το 1991 όταν το Ιράκ ε, εισέβαλε στο Κουβέιτ και δεύτερον όταν ε, υπήρξε ο τυφώνας Κατρίνα στον κόλπο του Μεξικού όπου ε, δίναμε 30.000 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα επί 30 ημέρες. Αυτός είναι ο στόχος και η αποστολή μας αλλά η αποστολή αυτή έχει διευρυνθεί τον τελευταίο καιρό διότι για να αυξήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο από πλευράς ε, του ο, πετρελαίου και του αερίου γιατί ξέρουμε ότι πολλές ε, ε, ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν για ε, ε, ε, για την ασφάλεια παροχής αερίου ιδίως με τους άγριους σημώνες που είχαμε το 2006 και το 2009 και η παροχή του αερίου συνεπιφέρει και κινδύνους για την ενεργειακή παροχή και όλα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε ε, την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα μειώνοντας ε, την κατανάλωση. Γιατί έτσι θα αυξήσουμε την ασφάλεια την ενεργειακή, αλλά γι' αυτό χρειάζονται ενέργειες για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα λόγω ιδίως των κλιματολογικών αλλαγών. Διότι αν δεν χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και να βελτιώσουμε ε, την εικόνα από πλευράς κυμνατολογικών αλλαγών. Οι προβλέψεις μας λοιπόν για τα θέματα της αποδοτικότητας του κλίματος και της ενεργειακής ασφάλειας, ε, τα δύο αυτά θέματα, οι κλιματολογικές αλλαγές και η ανάταξή τους και η ενεργειακή ασφάλεια είναι οι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος και ε, θέλω να σας πω πού έχουμε φτάσει και πού θα πάμε από εδώ και μπρο στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Καταρχήν θα ήθελα να σας δείξω έναν χάρτη ο οποίος δείχνει την ενεργειακή ζήτηση από τώρα μέχρι το 2030 και αφού ε, ξεπεράσουμε την ενεργειακή κρίση θα ξεκινήσει πάλι ε, την ε, οικονομική κρίση θα χρειαστεί το 2010 να υπάρξει μια ανάπτυξη της καταναλώσεως ενεργείας και θα φτάσει στο 22% το 2030 αν δεν ληφθούν από τις κυβερνήσεις πολύ σοβαρά μέτρα. Αυτό είναι το σενάριο αν όλα συνεχίσουν ως έχει κατάσταση, business as usual. Και βλέπετε ότι η αύξηση μπορεί να προέρθει από τον άνθρακα και δεν είναι ε, ένα παραδεκτό σενάριο από πλευράς ε, των κλιματολογικών αλλαγών. Σας δείχνω λοιπόν ε, μία διαφάνεια ε, ε, για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να συνεχίσει και να είναι ανεκτή αυτή η πρόοδος διότι εδώ βλέπουμε ε, την αύξηση που προβλέπεται σύμφωνα με τα διάφορα σενάρια. Βλέπετε λοιπόν ότι το σκούρο μπλε τμήμα είναι η παραγωγή από τα υπάρχοντα, τις υπάρχουσες πετρελοπηγές οι οποίες μειώνονται ταχύτατα ε, λόγω της ε, αφεμάξεως η οποία οφείλεται στη, φυσική, ε, στη φύση των πετρελαιοπηγών. Ε, υπάρχει ε, για να μπορέσουμε λοιπόν να αντεπεξέλθουμε θα χρειαστούμε το αντίστοιχο των 43 δισεκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που είναι τέσσερις φορές η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας για να ε, αντισταθμίσουμε τη μείωση. Οπότε έχουμε από τη μία πλευρά αύξηση της ζητήσεως, μείωση των πετρελαιοπηγών και άρα θα χρειαστούμε έξι Σαουδικές Αραβίες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν για να ε, ε, υπάρχει η παροχή του πετρελαίου που θέλουμε. Μετά υπάρχει το αέριο και εδώ τα ίδια διότι η ζήτηση του αερίου θα αυξηθεί διότι ε, είναι λιγότερο σημαντική για το διοξίσιο του ο άνθρακος η χρήση του αλλά και πάλι θα γίνουν τα ίδια. Δηλαδή η παραγωγή των υπαρχόντων πηγών θα μειωθούν όπως βλέπετε στο μοβ κομμάτι και ε, θα πρέπει συγχρόνως να αντισταθμίσουμε την αύξηση. Οπότε θα χρειαστούμε ε, επιπρόσθετα 2.500 TCM, δηλαδή τέσσερις Ρωσίες για να μπορέσουμε τέσσερις φορές την παραγωγή της Ρωσίας για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Οπότε ε, ε, υπάρχει το επιχείρημα ότι έχουμε πολλά αποθέματα ε, στο υπέδαφος αλλά θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις για να τα αξιοποιήσουμε στο μέλλον και από πλευράς κλιματολογικών αλλαγών και από πλευράς ασφαλείας είναι σοβαρά θέματα. Εδώ βλέπουμε εδώ τις εκπομπές του ενεργειακού τομέα. Οι αριθμοί οι οποίοι βλέπετε είναι κάπως χαμηλότεροι από το σύνολο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, αλλά αυτές είναι οι εκπομπές και μόνο. Και βλέπετε ε, ε, το πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο προέρχεται από τον ενεργειακό τομέα, άρα δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα. Η αύξηση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος σε διαφορετικά σενάρια προέρχεται από χώρες εκτός του ΩΣΑ, από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες και το πράσινο μέρος είναι το, η ε, ε, καύση του άνθρακα εκτός ΩΣΑ στην Κίνα που δημιουργεί τεράστιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Εάν λοιπόν υπάρχει μία πολύ σημαντική τεχνολογική διέξοδος για να μειωθεί η οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος είναι πώς θα τροφοδοτήσουμε ε, τους ε, ενεργειακούς σταθμούς ή στην Κίνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα για να μπορέσουμε να λύσουμε ε, το θέμα του διοξιδίου του άνθρακος. Λέμε ότι είναι μία δοκιμασία διαδικασία λίτμους ε, για να δούμε ε, ότι εάν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Και εδώ είναι η πρόταση ε, η οποία έχει διατυπωθεί για να μειώσουμε το θέμα των εκπομπών. Υπάρχει ένα σενάριο που οδηγεί σε, ε, ε, από 40 γιγατόνους σε 27, αλλά για να υπάρχει μία διαρκής εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση το ε, ε, έχουμε διατυπώσει ένα, ε, ένα πρότυπο για να μπορέσουμε να μειώσουμε κατά δύο βαθμούς και να, ε, και μειώσουμε στο ίμιση τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Πρέπει δηλαδή ε, να πέσουμε κάτω από το πράσινο και πρέπει να δούμε με ποια τεχνολογία θα γίνει αυτό. Τα περισσότερα, οι περισσότεροι πρόοδοι θα γίνουν σε χώρες εκτός του ΩΣΑ. Οι βόρειες χώρες και οι υποανάπτυξη χώρες θα χρειαστεί να πληρώσουν για ένα μέρος της ε, μειώσεως των χωρών του ΩΣΑ αλλά, ε, ε, εκτός ΩΣΑ αλλά είναι και αυτή μία λύση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Βλέπετε ότι το 2030 το 27% της μειώσεως θα γίνει με ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι ο όριμος καρπός που θα μπορέσουμε να, ε, να δεχτούμε. Και ε, έχουμε καταρχήν την Κίνα, έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας, μετά την ε, πυρηνική ενέργεια και το CCS κατά 10%. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και υπολογίζουμε και δείχνουμε στους διαπραγματευτές ε, σφαιρικούς αριθμούς αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η συμμετοχή κάθε χώρας ή κάθε περιοχής. Εδώ βλέπετε ότι το 2020, όχι το 2030, το 2020 ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη συμμετοχή θα είναι της Κίνας όπου υπάρχουν να μας δηλαδή εθνικά μέτρα τα οποία είναι ήδη εις το επίπεδο μειώσεως ενός γιγατόνου ή και περισσότερο το οποίο ε, είναι το 1 τέταρτο της αναγκαίας μειώσεως που χρειάζεται να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Λέγουν λοιπόν ότι δεν θέλουν να δεσμευτούν από πλευράς αριθμών αλλά να βελτιώσουν την ένταση ε, βελτιώνοντας κατά 40 ή 45% την επίδοσή τους. Αλλά ε, αν προσέξουμε μπορούν ε, να επιτύχουν κάτι καλύτερο, 47-48%. Η Κίνα έχει θέσει χαμηλούς στόχους, αλλά αν η Κίνα εφαρμόσει τα προγράμματά της και τις ενέργειές της αποτελεσματικά θα επιτύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Οι αριθμοί είναι σημαντικοί, αλλά βεβαίως τα μέτρα και οι ενέργειες είναι ακόμη πιο σημαντικές. Βλέπουμε ε, εδώ στην Ευρώπη μία μείωση κατά 0,4% γιγατόνων σε σχέση με τους στόχους για το 2000 30. Βλέπουμε ε, με βάση των αριθμών μία μείωση κατά 30% ε, σε σχέση με το 1990. Δηλαδή η δέσμευση της Ευρώπης για 20% είναι πολύ χαμηλή, αλλά πιστεύω ότι ρεαλιστικό επίπεδο είναι το 30%. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τώρα. Συγκρίνουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε και εδώ αναφερόμαστε σε μία μείωση 7-8% που είναι κάτι λιγότερο από ό,τι έχουν δεσμευτεί να κάνουν αλλά αν επιτύχουν αυτή την εσωτερική μείωση θα είναι σε καλό επίπεδο διότι οι αριθμοί της μειώσεώς τους είναι πολύ χαμηλοί και ε, από το ισχύον καθεστώς η μείωση θα, αυτή θα είναι σημαντική. Και εδώ είναι οι επιπτώσεις για ένα σενάριο για το, ε, για το σενάριο 450 όσον αφορά τις ενεργειακές ανάγκες. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες οι ενεργειακές καταναλώσεις θα φτάσουν στο νότερο σημείο ε, το 2020 και μετά θα αρχίσουν να μειώνονται. Ε, εάν λοιπόν λοιπόν ε, θέλουμε να πετύχουμε πρέπει τότε να έχουμε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και της ζητήσεως. Ε, ε, δεν πρόκειται για αύξηση της προσφοράς, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο υψηλότερο σημείο της ζητήσεως. Δηλαδή, ε, για να, υπάρχουν για υπάρχει μηδενικό διοξίδιο του άνθρακος, θα πρέπει να φτάσουμε σε μία φθήνουσα πορεία. Αλλά ακόμη και αν εξηγήσω το σενάριο αυτό, το 68% της, ε, ε, ε, της ενεργείας το 2030 θα προέρχεται ουσιαστικά από ορυκτά καύσιμα και το 2030 ακόμη ό,τι και να κάνουμε θα βρισκόμαστε με ορυκτά καύσιμα και γι' αυτό οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές. Αυτή είναι η τιμή την οποία προβλέπουμε για το ακάθαρτο πετρέλαιο αν όντως ακολουθηθεί αυτή η πορεία. Δηλαδή ε, η πραγματική τιμή θα είναι στο επίπεδο του 2008 και ε, ε, θα πάει από θα δούμε ότι θα φτάσει είτε στα 180 δολάρια είτε ε, θα πάει στα 130 δολάρια. δολάρια. Εάν όμως ε, υπάρξει αυτή η τιμή ε, για τις εκπομπές και καθοριστεί ε, σε 50 δολάρια το τόνο διοξιδίου του άνθρακος ε, και μετά φτάσει στους 110 δολάρια το 2030 τότε ε, θα καλύψουμε από εκεί τα 40 δολάρια λοιπόν όποιο και να είναι το σενάριο αναφοράς θα δείξει ότι η τιμή του πετρελαίου θα είναι ούτως ή άλλως πολύ ψηλότερη. Δηλαδή ε, η εποχή της φθηνής ενέργειας έχει τελειώσει και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και τα προγράμματα των κυβερνήσεων θα πρέπει να βασιστούν σε αυτό το γεγονός το οποίο πρέπει να αποδεχθούμε διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την υλοποίηση του σεναρίου 450. Ε, ακόμη και αν έχουμε το πράσινο, δηλαδή το φυσικό αέριο για το σενάριο 450 στο 2030, βλέπουμε ότι η Ευρώπη, η οποία είναι πολύ φιλόδοξη, θα χρειαστεί περισσότερο αέριο. Βέβαια η ασφάλεια του αερίου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό ε, πράγμα για να αυξήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια είναι να μην καταναλώνουμε το αέριο, θα πρέπει να διατηρήσουμε το αέριο, να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας, να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενεργείας ή, ή ε, πυρηνική ενέργεια, να διαφοροποιήσουμε αναλύσουμε τις πηγές ε, που μας τροφοδοτούν, να μην εξαρτώμαστε τόσο από τη Ρωσία αλλά περισσότερο από την ε, Κασπία, από τη Μέση Ανατολή, από το ε, υγροποιημένο αέριο, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τον αγωγό Ναμπούκο και η Ευρώπη θα πρέπει να μιλά με μία μόνο φωνή. Αυτή είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την ε, ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη στηρίζουμε διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε ε, να βελτιώσουμε και τις ανανεώσιμες πηγές και την ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να, οθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση <coughs> οδηγήσει της, την ενεργειακή της πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Στο διάγραμμα αυτό βλέπετε πόσο χρειάζεται να αυξήσετε την, ε, ε, τις δυνατότητές σας, διότι το κόκκινο πρέπει να μειωθεί θα πρέπει να αυξήσουμε κάπως το αέριο και ε, να βελτιώσουμε τη βιομάζα, την πυρηνική ενέργεια και άλλες. <clears throat> Βλέπετε όμως πόσο δύσκολο είναι όλα αυτά. Βλέπετε ότι πρέπει να δημιουργούμε κάθε χρόνο να χτίζουμε 18 πυρνικούς σταθμούς. Ε, πολύ περισσότερους από ό,τι πράττουμε τώρα. 700 ε, ανεμομήλους. Ε, 94 ε, πυρηνικά ε, κέντρα κάθε χρόνο, δηλαδή θα πρέπει να επενδύσουμε σε τεράστιες υποδομές για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Αλλά το κέρδος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι αριστερά βλέπετε τις επενδύσεις. Πρέπει να, να επενδύσουμε 8,3 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030 αλλά θα εξοικονομήσετε 8,6 ε, εκατομμύρια ε, από το λογαριασμό. Και εάν δείτε τη διάρκεια ζωής των επενδύσεων αυτών το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο. Πώς λοιπόν θα χρηματοδοτηθεί αυτό μέσω των επενδύσεων είναι ένα πολύ βασικό θέμα πολιτικής. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη τι έγινε στην Κοπεχάγη και να το αξιολογήσουμε. Διότι στην Κοπεχάγη περιμέναμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία επιτύχαμε. Αλλά οι χώρες δεσμεύτηκαν και η δέσμευση ε, είναι ε, περί αυτού, όχι στο 450 ε, ppm αλλά στα 550 ppm, δηλαδή αύξηση τριών βαθμών. Μπορούμε να πούμε όμως ότι με τις δεσμεύσεις αυτές έχουμε φτάσει κατά δύο τρίτα προς το στόχο μας. Έχουμε ακόμη να διανύσουμε ένα τρίτο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για να επιτύχουμε αυτήν την μείωση. Οπότε χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα της Κοπενχάγης και τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν. Ε, επίσης, η τα τεχνολογικά σχέδια για τεχνολογίες ε, με χαμηλές εκπομπές ή στον ηλιακό τομέα και άλλους. Θα σας δείξω ορισμένα παραδείγματα των ε, χαρτών πορείας τους οποίους δημιουργούμε. Εδώ βλέπετε την προηγμένη μορφή και βλέπετε ότι ο όλα τα προηγμένα αυτοκίνητα ε, ε, δεν θα έχουμε πλέον πωλήσει νέων αυτοκινήτων διότι είτε θα έχουμε υβριδικά είτε ηλεκτρικά είτε ε, αυτοκίνητα με ηλιακή ενέργεια και όλα αυτά είναι ένας πολύ ε, επίδοξος και φιλόδοξος στόχος και πρέπει όμως να επιτευχθεί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο των 450 για να μπορέσει να υλοποιηθεί το σενάριο 450. Πάλι απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις και έρευνα και πρόθεση της τεχνολογίας. Εδώ έχετε το χάρτη πορείας CCS μου ζήτησαν να αναφέρω 10 ή 20 πιλωτικά προγράμματα ε, φέτος και ε, καταρτίζουμε τον κατάλογο αυτό αλλά το 2020 δεν χρειαζόμαστε 20 αλλά 100 προγράμματα το 2030 χρειαζόμαστε 850 προγράμματα και χρειαζόμαστε 3.400 προγράμματα το 2050 ώστε το CCS να υλοποιηθεί και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν στόχος και θα πρέπει να αποδεχθούμε πραγματικά το CCS ε, και αυτό θα πρέπει να συμβεί ιδίω στις τυποανάπτυξη χώρες. Δηλαδή ε, το, η πλειοψηφία, το 65% ε, των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να υλοποιηθούν στις υποανάπτυξη χώρες πέραν των αγωγών και των άλλων προγραμμάτων. Πώς θα γίνουν λοιπόν αυτά. Μία κυβερνητική πολιτική με ένα πρόγραμμα εκπομπών 50 ή 100 ευρώ ευρώ είναι απαραίτητη για να μπορέσουν αυτά να υλοποιηθούν. Εδώ βλέπετε ε, την ε, ιδέα ενός ε, πανμεσογειακού πλέγματος ε, πόλεων ε, με ε, ηλιακή ενέργεια. Βλέπετε ότι ε, ένα μεγάλο μέρος της, της ένα μέρος της παραγωγής ηλεκτρισμού το 2050, 11%, θα υπάρχει εδώ των οποίων 1,5% θα είναι ηλιακή ενέργεια. Πρέπει να προωθήσουμε την ιδέα αυτή. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ακόμη για ενεργειακή αποτελεσματικότητα να ενισχύσουμε την τεχνολογία περιορισμού των εκπομπών και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, πρέπει να βελτιώσουμε και την ε, ασφάλεια από πλευράς παροχής φυσικού αερίου και ε, να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική. Ε, ε, συνεργαζόμαστε με όλους σας με μεγάλη χαρά και εδώ σας παρουσιάζω μία τελευταία διαφάνεια που βλέπετε τις εκπομπές διοξιδίου του ανθρακός να κατακεφαλίνα επ Δηλαδή κατά κεφαλήν ε, στην οριζόντια πλευρά. Πώς λοιπόν θα αποδεσμεύσουμε την οικονομική ανάπτυξη από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, πώς θα απελευθερώσουμε από το διοξίδιο του άνθρακος στην ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, ηλεκτροδότηση με ε, νέες πηγές ε, ενεργείας και βλέπουμε ήδη αλλαγές και πιστεύουμε ότι ίσως βρισκόμαστε ήδη σε ένα ιστορικό μετέχμιο για μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Υπάρχει βέβαια μία ανασφάλεια και γι' αυτό οι αυξομοιώσεις των τιμών των καυσίμων αντικατοπτρίζουν αυτή την ανασφάλεια. Ουσιαστικά όμως η ανασφάλεια αυτή ε, μας προβληματίζει και μπορεί να είναι και καλό στοιχείο διότι ε, προσβλέπουμε στο μέλλον πρέπει να υπάρξει αυτή η αλλαγή και νομίζω ότι η Ευρώπη είναι ο ηγετικός χώρος προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία συζητήσεις στο μέλλον και ε, θα παραμείνω καλός εταίρος προς εσάς, εγώ και η οργάνωσή μου και ελπίζω θα έχουμε καλή συνεργασία και στο μέλλον και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο να κάνω αυτή την παρουσίαση. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνακα για την παρουσίαση σα τι ε, πληροφορίε που μας διαθέσατε. Θα δώσουμε τώρα την ευκαιρία στους συναδέλφου να υποβάλουν και Κυρία Δεκαστήγιο, παρακαλώ, ως πρώτη. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πολύ και τον Πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την παρουσία του εδώ σήμερα. Μας δώσατε μια διεξοδικότατη εικόνα και πάρα πολλές πληροφορίες για αυτά τα σενάρια το 450 και την προοπτική για το 2030. Η ερώτησή μου είναι η εξής και σχετίζεται και με τις ε, δράσεις ε, για την ε, καταπολέμηση αλλαγής του κλίματος και την διάσκεψη της Κοπενχάγης και το μέλλον της Κοπενχάγης. Στην Κοπενχάγη είναι προφανές ότι δεν καταλήξαμε σε συμφωνία τουλάχιστον προς την άγουσα την οποία ε, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει δεσμευτική διεθνή συμφωνία για μείωση των εκπομπών ε, οι οποίες θα είναι και αυτές δεσμευτικές. Αλλά όπως είπατε και εσείς υπάρχουν μια σειρά από συμφωνίες που ήταν ε, οι πιθανές συμφωνίες και από αυτή την πλευρά μπορούμε να πούμε ότι είναι ενδιαφέρουσες. Πολλές δράσεις θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και προσπαθούμε να αναπτύξουμε κάποιες δράσεις, όπως για παράδειγμα στην Ένωση Ασίας Ειρηνικού, στην εταιρική σχέση Ασίας Ειρηνικού και εκεί εστιάζουμε σε περιφερειακό, σε τομεακό επίπεδο από κάτω προς τα πάνω. Η Ιαπωνία έχει μακρά πείρα επί του θέματος αυτού και εξ όσων γνωρίζω εγώ, βοήθησε και ε, με την εμπειρία της στη μείωση των εκπομπών των βιομηχανών, τουλάχιστον των ε, ε, βιομηχανιών που είναι μεγάλη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό όμως είναι πάντα εκτός των διεθνών ε, σενάριων που ασχολούνται με το θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα τα όσα συζητά ο ΙΕ και οι διάφορες διεθνείς οργανώσεις και τα βήματα που αναλαμβάνουν. Για παράδειγμα, δεν ήσασταν παρόντες στην Κοπενχάγη. Η δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμφωνίες οι οποίες ε, θα συμπεριλαμβάνουν και τις ε, βιομηχανίες που εκπέμπουν ε, πολύ διοξίδιο του άνθρακο και είναι από αυτούς που ε, είναι υπεύθυνοι για τα πολύ υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίω, που είναι υπεύθυνοι για όλες τις χώρες τις οποίες ε, είναι κατεστημένες αυτές οι επιχειρήσεις. Ε, το να έχουμε μια τομιακή προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Τι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι απώλεια δυνατοτήτων. Έχουμε τη δυνατότητα να δρώσουμε και δεν περιλαμβάνεται αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή στο μέλλον της Κοπενχάγης. Το τι μπορούμε να κάνουμε μετά από την Κοπενχάγη και ε, τι μπορούμε να κάνουμε μετά τις συνεδρίες που θα γίνει στο Μεξικό στο τέλος ε, του έτους. Η κυρία Ματουρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ε, Πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τανάκα για την παρουσία του εδώ στην Επιτροπή μας και για αυτό το τόσο πλήρες και τόσο ενδιαφέρον πλαίσιο που μας έδωσε για το τι γίνεται με την ενέργεια παγκοσμίω. Εγώ δεν θα σταθώ σε πολλά πράγματα γιατί η παρουσίασή σας ήταν ε, πλήρης, πολύ σαφής και μας έδωσε και πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστούμε. Μία παρατήρηση μου φάνηκε να λέτε ότι πέραν των μεγάλων επενδύσεων, εσείς θεωρείτε ότι είναι βιώσιμος ο στόχος που έχει θέσει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 για το 2020, 20% μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ισχύει αυτό. Θα ήθελα απλώς ένα σχόλιο από πλευρά σας κύριε Τανάκα για το θέμα αυτό. Ο κύριος Σοντή. Euh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ από πλευρά τον ομιλητή για τις, ε, δύο, για τις πολλές πληροφορίες που μας έδωσε. Έχουμε ζήτημα αρμοδιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι αρμόδια για την οργάνωση της αγοράς, την ασφάλεια και την ασφαλή χρήση αφενός, αλλά και τα κράτη-μέλη από την άλλη είναι αυτά τα οποία αγοράζουν την ενέργεια. Θεωρείτε λοιπόν ότι αγορεύει η αγορά, οι κανόνε τη αγορά την ενέργεια, ποια είναι τα οράματά σα και πω ε, η πραγματικότητα στον πλανήτη αντικατοπτρίζει την... Ε, συνθήκε τη της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραδείγματι καταδικάσει έναν ε, Ευρωπαίο προμηθευτεί για καταχρηστική για κατάχρηση εκμετάλλευση θέση στη Βόρεια Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια διαδικασία αγορά φυσικού αερίου στην Κασπία θάλασσα, ε, στη ζώνη τη Κασπία. Πιστεύετε λοιπόν ότι αντικατοπτρίζεται πραγματικότητα, γιατί εμεί είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα κληθούμε ε, δυνάμει των αρμοδιοτήτων μα να λάβουμε τι τελικέ αποφάσει. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σα για την πυρηνική ενέργεια, η οποία προχωρεί από ό,τι φαίνεται σε συνενετική ρύθμιση, σε συνενετική μάλλον αποδοχή, διότι δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα μεν. Θετώ όμως το ζήτημα, κάποιοι μιλούν για απόβλητα, εγώ εφευρίσκω τη λέξη υποπροϊόντα που μάλλον είναι και πιο εύυχη ε, υποπροϊόντα λοιπόν της πυρηνικής ενέργειας με δύο επιλογές ανά τον κόσμο. Η, την Αμερικανική η οποία λέει επιλέγουμε τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση και τη Γαλλική η οποία προχωρεί στην ανακύκλωση των υποπροϊόντων της πυρηνικής ενέργειας. Θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να αναπτυχθούν κονδύλια ή ταμεία επιστημονικής έρευνας για την πυρηνική ενέργεια έτσι ώστε να προαχθεί η έννοια της ανακύκλησης και να φτάσει ενδεχομένω και στο 100%. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χίμπνας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι, με βλέπετε. Ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε τα διάφορα ζητήματα τα σχετικά με την ενέργεια. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε τόσο ε, διεξοδική ανάλυση της ε, κατάστασης και με την ε, προσωμείωση των αναγκών μας σε ενέργεια και τις προτεραιότητες τις οποίες, οι οποίες μας αφορούν όλους και θα μας αφορούν και για το μέλλον μας μιλήσετε για διαφορετικές εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής και ε, τις ε, προσωμιώσεις που οδηγούν σε αυτές. Είπατε ότι υπάρχουν διαφορετικές τιμές και διαφορετικές προσωμιώσεις προς την τιμή. Επίσης, ξέρουμε ότι οι πολίτες ενδέχεται να αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο, φέρει πύρη, ενδέχεται να μην αποδεχθούν κάποιες τιμές. Φερρυπίν, το κόστος της ηλιακής ενέργειας ή της αιωλικής. Έχετε κάποια πρόταση έτσι ώστε να ενσωματωθεί, μάλλον να εξομοιωθεί σε όλη την Ευρώπη το κόστος ε, της ενέργειας, έτσι ώστε να μην πληρώνουν κάποιοι τα διπλάσια στη μια περιοχή από τη κάποια άλλη γιατί χωρίς ε, ομοιογενείς τιμές δεν θα είναι αποδεκτές, ε, αποδεκτές από τον πολίτη προτάσεις. Για την ε, κύρα που μας είπατε ότι είναι ο δεύτερος την τάξη, έχει τις δεύτερες εκπο, σε μέγεθος εκπομπές στον κόσμο. Πώς μπορούμε να πείσουμε την Κίνα να ακολουθήσει, να εισαγάγει στις μεθόδους παραγωγής της τη σύγχρονη τεχνολογία. έτσι ώστε να ε, βελτιωθεί το επίπεδο των εκπομπών της κυρία Καρβάγιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Τανάκα. Ήταν όντως πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όσους καλούνται να λάβουν τις αποφάσεις. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις για το CES. Είπατε στο σενάριό σας ή τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα προκαλούνται στο μεγιστό τους ε, βαθμό, στο μεγαλύτερο του ποσοστό από χώρε έξω από τον ΩΣΑ. Είπατε ότι έχουν μεγάλη σημασία για την Κίνα. Είπατε επίσης, ε, μίλησατε για το σενάριο 450 και τη δυνατότητα περιορισμού των εκπομπών μόνο κατά 10% ανά τον κόσμο. Γιατί δεν είναι επαρκή η, ε, η τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της αποθήκευσης, της σύλληψης και αποθήκευσης ε, διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, για μια εικόνα της Ευρώπης το 2020, ε, ασφαλώς το φυσικό αέριο θα είναι θεμελιώδη σημασία για την Ευρώπη. Όμω χρειάζεται η διαφοροποίηση εξαρπαντό. Και ρωτώ εάν συμφωνείτε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας κεντρικός αγωγός όλη την Ευρώπη για το υγραέριο, για το υγροποιημένο μάλλον φυσικό αέριο. Βλέπω όμως από, τη γεωγραφική, από την εικόνα τη γεωγραφική που μας δίνεται ότι δεν ε, ε, προτείνεται την, απόλυ, την ε, εκτεταμένη χρήση του και μεταφορά του πάνω απ' όλα δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει σημαντικό ρόλο ενώπιση και τη διαφοροποίηση στην Ευρώπη. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Κύριο Στανάκα, για να απαντήσει παρακαλώ σε αυτόν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ήταν πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Τομεακές προσεγγίσεις από τη βάση προς τα άνω. Όταν υπολογίσουμε, και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα από τα προσαρτήματα στα γραφήματά μας, ε, εάν υπολογίσουμε αυτό το σενάριο του 450, το όντι, είναι πρακτική η προσέγγιση που επιλέγουμε, υπάρχουν τομεακές προσεγγίσεις γίνεται λόγος για κάποιες τομεακές προσεγγίσεις και συμφωνίες. Ας δούμε λοιπόν αυτές. Ας δούμε πρώτα τις κύριες, τους κύριους τομείς εθνικό επίπεδο τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη με τις εθνικές πολιτικές και την τομεακή μεταπροσέγγιση, την οποία την έχουμε είτε για, το, για τη χαλιβουργία, είτε για την τσιμετοβιομηχανία, την αεροναυπηγική, τις μεταφορές, το τομέα του σιδήρου, με τα πιο αποτελεσματικά πρότυπα ε, και κάνουμε προβολή του εάν υπάρξουν κάποιες συμφωνίες προς την τάδε κατεύθυνση, τι είδους μειώσεις σε εκπομπές μπορούμε να περιμένουμε. Ένα γιγατόνο είναι η απάντηση, αλλά πάλι χρειάζεται η μείωση κατά 1,8 γιγατόνους στο 2020. Επομένω, και αν δούμε ακόμα τις χώρες του ΩΣΑ ως μία ενιαία αγορά, θα πρέπει να δούμε τι είδους μηχανισμούς ανώτατων ορίων και ε, ανταλλαγής μπορούμε να προβλέψουμε. Για το 2020 προβλέπεται περίπου 50 δολάρια ένα τόνο του διοξιδίου του άνθρακα με αυτή την ε, προβολή μας. Προσπαθούμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο πρακτική προσέγγιση, πιο ρεαλιστική προσέγγιση με ένα μηχανισμό cap and trade ε, ενιαίο στον κόσμο, ασφαλώς δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Θα είναι ίσως πιο αποτελεσματικός ως προς τη χρήση ενέργειας τρόπος για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συμβεί ε, υπ' αυτούς τους όρους. Ε, απλώς το κοιτάμε ως ιδεώδη στόχο και προσπαθούμε να δείξουμε ότι ο συνδυασμός τέτοιων ρεαλιστικών μέτρων μπορεί να μας, μπορεί να μας οδηγήσει στο σενάριο 350 Και έτσι έχουμε με ε, με αυτή την προβολή το 2020 το 2020 50, ε, τόνους, 50 δολάρια ανά γιγατόνο και 150 για το 2030. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε μια συγκράτηση στο 2020 και μετά στα, ε, ριζική, ραγδαία μείωση. Το 2020 με την προβολή αυτή είναι εφικτός στόχος, αλλά πρέπει να είναι πολύ ψηλή, όπως είπα, η τιμή ανατόνο. 50 δολάρια, όπως είπα, για να έχουμε τους στόχους του 2020 προς την αποτελεσματικότητα και τη μείωση των εκπομπών του του άνθρακα ή, την, ή το μείγμα των ανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως προς το ζήτημα των αγορών στην Ευρώπη, και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ε, ζήτημα, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η ενέργεια στην ασφάλεια πρέπει να έχει μια συνιστόσα ασφάλειας της αγοράς. Δηλαδή με την πιο αποτελεσματική χρήση, αποτελεσματική χρήση δηλαδή, της ενέργειας και προσέγγιση αγοράς. Αυτός είναι ο συνδυασμός. Και τρίτον, για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ενιαία αγορά για την ενέργεια. Αυτή είναι η ιδεώδης επιλογή. Και πάλι υπάρχουν στοιχεία με πολύ καλά παραδείγματα από τα σκανδιναβικά κράτη για τα λεγόμενα pools, για την κοινή χρήση δηλαδή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ισπανία με την Πορτογαλία επίσης έχουν αναπτύξει την αγορά τους ε, στην Ιβηρική Χερσόνεξο, πάλι για την ηλεκτρική ενέργεια. Και μας δείχνουν αυτά τα παραδείγματα ότι μία ενιαία αγορά ενέργειας με καλή διασύνδεση μεταξύ των κρατών, πέραν των σύνορων δηλαδή, ή ένα δίκτυο για το φυσικό αέριο πέραν των σύνορων, και εάν υπάρχει εναρμόνιση των κανόνων, των ε, ρυθμίσεων ή μια, μια ενιαία υπηρεσία ρύθμισης της αγοράς ενέργειας, γιατί βέβαια χρειάζεται ρύθμιση στην αγορά, αλλά βέβαια Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί και η ασφάλεια και η χρήση τη ανανεώσιμων πηγών ενέργεια για το μέλλον. Πυρηνική ενέργεια. Ναι, το όντι. Ο πρόεδρος σας, ο κύριος Μπαρόσο, από ό,τι μάθαμε, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα μόλις μια σαφέστατη δήλωση στο Παρίσι. Μάλιστα, εγώ ήμουν και παρόν. Με εντυπωσίασε, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ιστορική μεταστροφή της πολιτικής Ευρώπης σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Ασφαλώς, βέβαια, Πρόκειται για μια ε, πηγή ενέργειας χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα με μεγάλη σημασία για την λύση των προβλημάτων σε όλο τον πλανήτη. Δεν αποτελεί τη μοναδική λύση, αλλά αποτελεί σημαντικό τμήμα της λύσης για όλο τον πλανήτη. Έτσι πιστεύουμε εμείς. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αποβλήτων, το όντι, είτε με την ε, ε, επανεπεξεργασία ε, και νέα χρήση. Υπάρχουν διαφορετικές λύσεις που έχουν επιλέξει διάφορε χώρε, Δύσκολο ζήτημα, πολύ σημαντικό ζήτημα. Αλλά ακόμη και με τη διαχείριση των αποβλήτων έχουμε νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον γράφωμα εδώ του κόστους ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο θα δείτε την επόμενη εβδομάδα. Είναι μια δημοσίευση η οποία δεν έχει ακόμη ε, διατεθεί στο κοινό. Από αυτό όμως το γράφημα βλέπετε ότι έχουμε 30 δολάρια ανατόνα δεξιδίου του άνθρακα με σαφή απόδειξη του γεγονότος ότι η πυρηνική ενέργεια συγκρινόμενη με άλλες πηγές είναι μια φθηνή επιλογή. Με καλή σχέση κόστος αποτελέσματος δηλαδή. Εάν επομένως επιλέξει κανείς σε μια χώρα αυτή την ε, επιλογή, το όντι, την συνιστούμε και εμείς. Πρόκειται για ένα αναγκαίο τμήμα μια λύση. Αλλά ταυτόχρονα υπό τον όρο ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι όροι της ασφάλειας, της ακίνδυνης χρήσης και της μη διάδοσης. Ξέρουμε ότι είναι πολλές οι χώρες που τώρα, ε, από τον τρίτο κόσμο που τώρα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια. Πρέπει οι ίδιοι κανόνες με κάποιο τρόπο να επιβληθούν σε διεθνέ επίπεδο και σε αυτέ τι χώρε ασφαλώ. Και για να περάσω στην τέταρτη ερώτηση για την ε, αγορά, την γλυακή και αιωλική ενέργεια και την εναρμόνιση, την οποία αναφερθήκατε. Βεβαίω και συμφωνώ, όμω σημαντικό είναι ότι και η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, οι ανανεώσιμε πηγέ δηλαδή, χρειάζονται κάποια υποστήριξη από τι κυβερνήσει, γιατί χωρί αυτήν δεν μπορεί καν να ξεκινήσει, να γίνει η εισαγωγή τους ε, στο ενεργειακό μείγμα. Χρειάζεται όμως μια προβλέψιμη πολιτική, κρατική πολιτική για το μέλλον. Εάν δεν γνωρίζουμε ποιε θα είναι, είναι οι τιμέ στο μέλλον για την ε, ενέργεια, ε, δεν θα επενδύσει ο ιδιωτικό τομέα. Άρα χρειάζονται κάποιε ενδείξει για το προ τα που πηγαίνει η αγορά, ποιε θα είναι οι συνθήκε. Και επίση χρειάζεται και μία σταδιακή κατάργηση των ανεσχήσεων, των, στήριξη δηλαδή από τι κυβερνήσει, όταν θα είναι όριμε οι συνθήκες βέβαια, σταδιακή. Έτσι ώστε εν τέλει και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση των τιμών στι διάφορε χώρε από την αγορά, από πλευρά τη αγορά. Η Κίνα χρειάζεται δυστυχώς το σύστημα της ε, σύλληψης και αποθήκευσης άνθρακα ε, θα πρέπει η, του, η Κίνα να περάσει το σύστημα cap and trade οπωσδήποτε. Έχει ένα υψηλό κόστος ασφαλώς. Μια άλλη λύση είναι το CCS να μπει στον ε, μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης, δηλαδή να χορηγηθούν πιστώσεις για την ανάπτυξη του CCS. Υπάρχει δηλαδή ε, η ένδειξη ότι δεν μπορεί το CCS να ε, απογειωθεί, θα έλεγα, εάν δεν υπάρξει κάποια υποστήριξη με επιδοτήσεις. Επίσης, το 10% της έκπτωσης πρόκειται από το CCS. Για να μπορέσει στην πράξη να εφαρμοστεί το σύστημα σύλληψης και αποθήκευσης. Ε, για το 2020. Αλλά όπως είπα, για να απογειωθεί αυτή η τεχνολογία πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος, να εγκριθεί από τα κράτη του ΟΣΑ, και μετά να προχωρήσει πάνω απ' όλα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως ε, της Κίνας, έτσι στο 2030 να είναι, ίσως όχι σε εμπορικό επίπεδο, αλλά να έχει ξεκινήσει σε να αποδεικνύει την εμπορική του χρησιμότητα, αλλά πάντοτε θα είναι σε απόλυτη ανάπτυξη την εποχή εκείνη. Το 2050 όμως πιστεύουμε ότι από όλη την... Ε, ε, από όλο το μείγμα παραγωγής ενέργειας θα έχουμε τις ανανεώσιμες, πηγές κατά 50% και κατά 50% την πυρηνική ή το CCS. Θα δούμε το μείγμα πώς θα προσχωρήσει. Η διαφοροποίηση στο, φυσικό, στο αέριο στην Ευρώπη ναι, είναι πολύ σημαντική. Ε, δεν φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στο, τμή, στο, στο δικό μου γράφημα, αλλά έχουμε μέσω πρόθεσμα το υγροποιημένο αέριο, το οποίο δεν έχει προχωρήσει τόσο ε, στην Ευρώπη, περισσότερο σε άλλες χώρες, αλλά πάντως λόγω της έντασης εκπομπών του άνθρακα θα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο αέριο. Το υγροποιημένο είναι φυσικά πολύ σημαντικό και για λόγους ασφάλειας των προμηθειών της, της χρήσης ενέργειας. Γνωρίζουμε ήδη ότι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν ξεκινήσει εγκαταστάσεις για το... έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται εγκαταστάσεις για το υδροποιημένο φυσικό αέριο και νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ως προς την προμήθεια της Ευρώπης σε ενέργεια. Ο Πρόεδρος. Κύριε Τάνακα, σας ευχαριστώ θερμά. Πολλές φορές υπάρχουν ε, εκδηλώσεις ή συναντήσεις και πολιτικές συζητήσεις και ε, λέει κανείς ε, είμαι ευτυχής που ήμουν εδώ και κρίμας που δεν ήταν και περισσότεροι διότι για τα θέματα ασφαλείας όπως και για το θέμα το πώς μπορούμε να απαντήσουμε επικοδομητικά στο θέμα της ενεργειακής ασφαλείας δεν φτάνει κανείς να πιστεύει και να ονειρεύεται αλλά χρειάζονται ε, αριθμοί και δεδομένα και σας ευχαριστώ διότι μας βοηθήσατε να συγκεντρώσουμε ορισμένα στοιχεία. Όχι δηλαδή ενδεχομένως όλη την αλήθεια αλλά και αυτό μπορεί να βοηθήσει και θα βοηθήσει διότι θα μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συζήτηση μεταξύ μας γιατί είναι δύσκολο. Όποια και να είναι η πολιτική τοποθέτηση πρέπει να υπάρξει μια αντικειμενική συζήτηση επιβάσει απόψεων ξύπνων ε, από ε, ε, στοιχείων λογικών δαπανών για να ξέρει κανείς που πάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ διότι σε πολλά σημεία, όχι μόνο σε ένα, μας, μας εξυπηρετήσατε πολύ, μας ανοίξατε τα μάτια και πρέπει να σας πω ότι οι εκδηλώσεις όπου ανοίγει το μυαλό και που αρχίζει κανείς να αναρωτιέται είναι οι καλύτερες Γι' αυτό και σας ευχαριστώ ακόμη και αν αργά το απόγευμα είχαμε τη δυνατότητα να σας συναντήσουμε και σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συνάντηση.